Να ακούσουμε τις ερωτήσεις από πλευράς των μελών τώρα. Έξι άτομα έχω ζητήσει το λόγο. Να ακούσουμε λοιπόν όλους τους βουλευτές και στη συνέχεια να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Να σας πω ότι είναι περιορισμένο το χρονοδιάγραμμα. Αρχικά προβλεπόταν μόνο μέχρι τις 15 και 40 το θέμα αυτό. Δεν θα προλάβουμε βέβαια αλλά, εν πάση περιπτώσει, φροντίστε να είναι συντόμε οι ερωτήσει σα. Η κυρία Ρέντα είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την επισκόπηση που μας έδωσε. Θα ήθελα να σας πω ότι θέλω να μας πείτε ποια θα είναι τα θέματα τα οποία θέλετε να τονίσουμε στο μέλλον. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ, πριν από κάποιους μήνες ανακοίνωσε στην Επιτροπή τάξη και μάλιστα το επανέλαβε πρόσφατο σε μια συνέντευξη ε, στην Le Monde ότι θα ήταν υπέρ μια νομοθεσία υπέρ τη προστασία των πληροφοριοδοτών, των whistleblowers. Και όντω έχει ζητηθεί να κατευθυνθεί τέτοια πρόταση μέχρι τον Ιούνιο. Αλλά έχουμε φτάσει πλέον Ιούνιο. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει παρουσιαστεί τέτοια έχει δημοσιευτεί τέτοια πρόταση οδηγίας μέχρι το Μάιο για την προστασία των ατόμων αυτών. Νομίζω ότι πολλές ε, ομάδες στο Κοινοβούλιο θα ήθελαν να υπάρξει μια κινητοποίηση προς την κατεύθυνση αυτής. Πώς θα το καλύψετε λοιπόν το θέμα της ε, προστασίας των πληροφοριδιωτών. Νομίζω ότι θα αποτελούσε αυτό μια καλή αντίδραση και στα έγγραφα του Παναμά, όχι μόνο τα θέματα τη περιεχομένου, αλλά και το θέμα της προστασίας των πληροφοριοδοτών. κυρία Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Νομίζω ότι μας δώσατε μια πολύ καλή επισκόπηση της κατάστασης. Τρία σημεία θέλω να δείξω. Καταρχάς, την προηγούμενη Τετάρτη και Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε ένα ψήφισμα με μια έτοιμη πρόταση μάλιστα για μια ανοιχτή, αποτελεσματική και διαφανή διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματο όλη τη Επιτροπή και σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου, ότι είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι από την ψυχρή αντίδραση του Αντιπρόεδρου Κατάινεν και όλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι κρύφτηκε πίσω από τη δικαιολογία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ήδη πολλά για την καλή και σωστή διακυβέρνηση και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί με το one size fits all. Λες και εμείς ζητάμε για κάτι ενιαίο, κάτι το οποίο θα εναρμονίσει και θα κωδικοποιήσει όλα τα στοιχεία που δεν υπάγονται στις βασικές αρχές της καλής διαχείρισης, καλής διακυβέρνησης. Σας ερωτώ λοιπόν, ως Επιτροπός Αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, προτίθεστε να προωθήσετε το σχέδιο κανονισμού, το σχέδιο νομοθεσία αυτή και να συνεργαστείτε με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν και την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα που έχει αρμοδιότητα. Κατά δεύτερον, αναφέρατε, για τις, δύο προτάσεις για τις ε, συμβάσεις online. Και χαίρομαι που θέλετε να γίνει η δουλειά αυτή εκ παραλλήλου. Τι γίνεται όμως με το refit της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση για τα απτά αγαθά. Ελπίζω να μην καθυστερήσει η δουλειά αυτή. Τρίτον, εν συντομία πάλι, να σας ευχαριστήσω όλο ιδιαίτερος για την ε, πρόθυμη συνεργασία με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, παροχή αγωγής ε, των χωρών, των συνδεδεμένων χωρών σε θέματα δικαιοσύνης. Ελπίζω λοιπόν να είναι αύριο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 είχαμε ζητήσει να υπάρχουν συγκεκριμένες αποζημιώσεις ε, προκαταβολικά ε, για να μπορούν να καλυφθούν όλοι όσοι χρειάζεται να αποζημιωθούν. Δεν υπήρξε καμία λύση εκτός από ένα εκτιμώντα από το οποίο παρέπεμπε την επίλυση του προβλήματος σε κάτι άλλο, ή στην οδηγία δηλαδή και στην ανασύνταξη η ενωθέρωση αυτής. Επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο ήθελα να ρωτήσω εάν το θέμα των ε, όρων των συνθηκών εργασία των εξαρτάμενων εργαζομένων θα εξεταστεί, όπως είχαμε πει ότι θα γίνει. Ε, Mr. Ε, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλή επισκόπηση. Τρία σημεία να αναφέρω αφενός σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την αγορά αγαθών. Να φροντίσουμε προκειμένου να μην υπάρξει πολυτερόκλητη εικόνα πολλά ετερόκλητα στοιχεία σε ό,τι αφορά την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο, σε ό,τι αφορά τις ε, εξαποστάσεως πωλήσει και την οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά. Τρία διαφορετικά νομοθετήματα ε, θα έχουμε, όπου νομικός πώς θα πρέπει να υπάρχει και μια ομοιογένεια, να μην υπάρξει κατακαιρματισμό σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση και των σχετικών ε, συμβάσεων να το έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη. Ιδιαίτερα γιατί ως ε, επιχειρήσεις δεν είμαστε B2B, δηλαδή δεν είναι μεταξύ επιχειρήσεων οι πωλήσει, αλλά B2C μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτή. Να μην υπάρξει υπερβολικό κατακριματισμό και υπερβολικά περίπλοκη διαμόρφωση τη νομοθεσία σε ό,τι παρά τι μονοπρόσωπε εταιρείε. Ένστικτο πώ θα έλεγα ότι έτσι όπως έχει πρόταση δεν θα συγκεντρώσει πλειοψηφία. Καλά θα ήταν να βρούμε λοιπόν, θεωρώ, ένα δρόμο και αυτό με συνετικό τρόπο μάλιστα, προκειμένου αυτά που είναι θετικά και καλά να μπορέσουμε να τα προαγάγουμε και αυτά που μας προβληματίζουν σε ό,τι αφορά τη διάσταση να αποκλειστούν για να διαμορφωθεί μια σωστή πλειοψηφία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε ένα εταιρικό δίκαιο, μια διαμόρφωση της εταιρικής νομοθεσίας να παρέχουμε ως νομοθέτες. Και γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να κάτσουμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα επί της αρχής και να ακολουθήσουμε και μια πιο συνενετική μορφή η οποία θα αποκλείσει, αν θέλετε, τις αμφιβολίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή και ίσως να το δώσουμε και ένα περιεχόμενο το οποίο θα μας καλύψει. Τρίτο σημείο. Μιας και μιλήσατε για τις επιχειρήσεις και πώς μπορούν να είναι έτοιμες για την ψηφιακή αγορά. Έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία είναι ευκταία στο σημείο αυτό. Ε, είμαστε στην εποχή, ξέρετε, στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Θα υπάρχουν πολλές διαδικασίες αυτοματοποιημένες και αυτό αποτελεί ένα βήμα όπου θα ξεπεράσουμε το εταιρικό δίκαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διάφορα στοιχεία θα γίνονται μηχανικά. Θα θέλαμε λοιπόν να σας προτείνουμε πρόταση η οποία θα ρυθμίζει το πώς θα α, ρυθμίζονται τα πράγματα μεταξύ των συσκευών, μεταξύ των μηχανών. Επίσης, σε διάφορες περιστάσεις ακούω την ιδέα και την έννοια της ιδιοκτησίας των δεδομένων. Από νομικής άποψης δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, αλλά εκ πρώτης όψεως θα έλεγα ότι αν περάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αν θελήσουμε να ρυθμίσουμε και τις μικρότερες και τις πιο ε, επουσιώδεις λεπτομέρειες για την ιδιοκτησία των δεδομένων, δεν θα βγάλουμε άκρη. Θεωρώ ότι ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλα μοντέλα, πώς θα υπαχθούν όλα αυτά σε μια ε, διαφανή νομοθεσία και ρύθμιση. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σε κλειστά συστήματα ενδεχομένω. Αυτό να έχει νόημα. Αλλά σε ανοιχτά συστήματα θεωρώ ότι χάνουμε σε ό,τι αφορά το θέμα της ιδιοκτησίας και θεωρώ ότι ο αστικός κώδικας ολόκληρος θα μπορούσε να ασχολείται μόνο για τα δεδομένα. Αυτό το αναφέρω μόνο και μόνο για να σας πω ότι θα πρέπει να ρωτηθούμε κατά πόσο έχει νόημα καν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. προτού όλα αυτά πάρουν διαστάσει που δεν θα επιτρέπουν πλέον να τα εντάξουμε σε ένα μόνο πλαίσιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την πολύ συνοπτική σα παρουσίαση. Έχω διάφορε ερωτήσει να θέσω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τι ε, διαδικασίε χρεοκοπία αφρεγγιότητας οι ιδιωτικέ ε, τέτοιε διαδικασίε λαμβάνονται υπόψη, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχει χάσει τα σπίτια του. Η Επιτροπή ε, έχει σκεφτεί το θέμα τη προσωπική χρεοκοπία. Κατά δεύτερον, Women on Board. είπετε από 10 μέχρι 21%. Βλέπουμε λοιπόν ε, ότι υπάρχει αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, αλλά αυτό συμβαίνει εκεί που έχουν βρεθεί εθνικές λύσεις αντιμετώπισης του θέματος και ξέρω ότι τον ίδιο σκοπό επιδιωκούμε στο θέμα αυτό. Ερωτώ λοιπόν, τι σημαίνει αυτό από πλευρά δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Πανελέκτη, ότι αυτό το θέμα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Βρυξέλλες 2α. Το επόμενο θέμα μου λαμβάνεται υπόψη τις ελάχιστες ε, προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα παιδιά, για παράδειγμα, να υπάρχουν δηλαδή κάποιες ε, σε ό,τι αφορά τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες διαφορές και χρειάζεται μια ομοιογενοποίηση. Και τέλος, η εταιρεία ε, με ένα μέλος μόνο. Στην προ... παρουσίασή σας Αναφέρατε διάφορα στοιχεία, υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση σας ό,τι αφορά τα έγγραφα του Παναμά. Δεν θα αφιστεί διαφάνεια και σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά μητρώα. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι υποχρεωτικά αυτά και θα πρέπει να ενημερωθούν, παρόλα αυτά να ενημερωθούν σε άλλες χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εντελώ διακοσμητικά. Είναι πολύ διαφορετικά λοιπόν τα πρότυπα. Και άρα πώς μιλάμε για πλήρη διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη μάλλον τα, τα αντιλαμβάνεστε αυτά και δεδομένων όλα αυτά των δεδομένων Μήπως θα αποσύρετε την, την πρότασή σας και σε ό,τι αφορά και την 14η ε, οδηγία για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισκόπηση αυτή που μας δώσατε. Τρία σημεία θέλω να θίξω. Τα πρώτα δύο είναι νομικά ζητήματα για την ε, Συμφωνία Ελευθεροπορίου ΣΕΤΑ για τη σύσταση ε, δικαστηρίων διαιτησίας που προβλέπονται tribunals, ε, δικαστήρια. Μεταξύ άλλων και για την προστασία την επενδυτική των επιχειρήσεων. Εδώ εκφράζονται αντιρρήσεις από πλευράς των ε, γερμανικών δικαστηρίων και από ευρωπαϊκές ενώσεις δικαστών σε ό,τι αφορά τα δικαστήρια αυτά τα οποία θεωρούνται ότι παραβιάζουν τη συνθήκη της Λισαβόνας ή θα παραβίασαν άμα συστήνονταν. Γιατί ουσιαστικά de jure, μάλλον de facto, όχι de jure αλλά de facto, ε, δημιουργείται ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα. Εκφράζονται λοιπόν βασικές αμφισβητήσεις του κράτους δικαίου, της νομιμότητας. Αυτό το επικρίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Δεύτερη ερώτηση για τη νομική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προορίζει την ΣΕΤΑ για ένα αμυγός ευρωπαϊκό επιχείρημα, μια ε, αμυγός ευρωπαϊκή σύμβαση. Συμφωνείτε, είναι αμυγός ευρωπαϊκή σύμβαση αυτή. Δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν καθόλου τα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή. Τρίτη ερώτηση. Η οδηγία για το εμπορικό απόρριτο, trade secrets, το οποίο αποφασίστηκε στο Κοινοβούλιο πριν από κάποια εβδομάδα, ο Σέντζιο Κονφεράτη, ε, πρότεινε και εφήρμοσε εκεί μια ιδιαίτερη προστασία των whistleblowers θα με ενδιαφέρει κατά πόσο μπορείτε να αναλάβετε την πρωτοβουλία προκειμένου να εφαρμόσετε αυτή την ιδιαίτερη προστασία των πληροφοριοδοτών. Γιατί θεωρώ ότι οι πληροφοριοδότε δεν είναι στοιχεία τα οποία είναι απολύτω απαραίτητα για τη διαφάνεια. Για τη φοροδιαφυγή και είναι μεγάλη η, η υπηρεσία που παρέχουν. Θα ήταν μεγάλη η υπηρεσία που παρέχετε και εσεί αν θα μπορούσατε να προστατεύσετε του whistleblowers. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα δίναμε μια μεγάλη υποστήριξη και στη δημοκρατία στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση από την ε, Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση για τους ευάλωτους ενήλικες που είναι ένας φάκελος τον οποίο ε, έχω αναλάβει κάποια καθήκοντα και θα ήθελα να πείτε πώς συνδυαζόμαστε εδώ με τη φιλοσοφία που έχουμε πάντα στην Ευρώπη. Θα πρέπει τους πιο εύθραυτους ανάμεσά μας να τους προστατεύουμε και να μην τους επιτρέπουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και νομίζω πως είπατε πως δεν είναι υπέρ αυτής της έκθεση η Κομισιόν για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να σε την προσοχή και νομίζω πως η εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν μας είπε πως έχει πολλούς δισταγμούς γιατί είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις όπου ε, υπάρχει ε, χρησιμο... χρειάζεται τη προστασία. Αλλά από το δικαστήριο της ε, ΛΙΛ μου είπαν πως υπάρχουν τουλάχιστον χίλιες υποθέσεις που περνάνε από τα δικά τους ε, δικαστήρια με θέματα κυδαιμονίας ατόμων ε, στην ευρύτερη περιοχή. Στο δε πολύ μικρό δικαστήριο της περιοχής Βαλενσίνη ήταν τουλάχιστον 400 αυτές οι υποθέσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι λίγα αυτά τα παραδείγματα και θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να το αντιμετωπίσετε με πιο θετικό πνεύμα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξατε και που αποτελούν κομμάτι της συζήτησής μας. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση του κ. Βλόν, γιατί καταλαβαίνω πως και για εσάς στην Επιτροπή Γιούρη είναι σημαντικό το θέμα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα συζητάμε ε, τις αρμοδιότητες, μια και πρόκειται για οριζόντιο θέμα που καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή γίνονται εντατικές συζητήσεις με τον συνάδελφο τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος μου ζήτησε να συμμετέχω πιο ενεργά στο θεματολόγιο κατά της διαφθοράς. Και νομίζω ότι εκεί ε, θα καλυφθεί το θέμα σας, αλλά υπάρχει ένα νομικό ζήτημα και θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ε, το θέμα αυτό να δρομολογηθεί για να λάβει συνέχεια. Και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που μας συζητάτε είναι μια πιο ολοκληρωμένη έκθεση για το πώς θα το ε, αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θα σας το φέρω ενδεχομένω στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε στην Επιτροπή που νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο. Δεν σχεδιάζω εγώ αυτές τις συνεδριάσεις, αλλά νομίζω ότι θα είναι μάλλον Σεπτέμβριο. Άκουσα μία ερώτηση για ανοιχτή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, ε, ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες που έχουμε, γιατί πρόκειται για αρμοδιότητες που μοιράζονται τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε υπέρ της εφαρμογής ε, μιας ε, ομάδας αρχών που θα επιβάλλονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σας πω πως και εγώ η ίδια έχω περάσει από όλε τι βαθμίδε τη ε, τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μου. Οπότε νομίζω ότι είμαι αρκετά καλά εξοπλισμένη σε προσωπικό επίπεδο για να αντιμετωπίσω το, τη συζήτηση του θέματο αυτού. Πρέπει όμω να δούμε τι γίνεται με τι αρμοδιότητες και να δούμε σε νομοθετικό επίπεδο αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους μέτρα. Έχει προσφερθεί πολύ χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη μέσω του ΕΚΤ για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και νομίζω πως ίσως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε Ποιε είναι οι αρχέ που θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν χρησιμοποιούν ε, κοινοτική χρηματοδότηση. Και ίσως αυτό να είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος για να το πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε νέα νομοθεσία, αλλά η νέα νομοθεσία πάντα χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ίσως λοιπόν... Αν το δούμε σε επίπεδο χρηματοδότησης έργων, να τα καταφέρουμε κάπως καλύτερα. για, τα, για τις ψηφιακές συμβάσεις Έχουμε ξεκαθαρίσει στο Συμβούλιο πως θέλουμε αυτό να αποτελέσει ένα πακέτο δύο προτάσεων. Κατανοούμε όμως πως υπάρχουν δύο διαφορετικές θέσεις στην νομοθεσία αυτή που έχουμε και την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο όπου εκεί ενδεχομένως η θέση είναι πιο ευνοϊκή μια και δεν υπάρχει τέτοιου είδους νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Δύο μονοκράτη μέλη έχουν δεταστήσει τέτοιου είδους νομοθεσία, οι κατοχώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε και την ενιαία ψηφιακή αγορά και το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελεί και το αγαθό το οποίο ε, με το οποίο συναλλασσόμαστε διασυνοριακά, καταλαβαίνετε πως υπάρχει ε, στήριξη από τα κράτη-μέλη για την οδηγία αυτή. Μια οδηγία που ασχολείται με τους συμβατικούς όρους και με το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποζημίωση για άτομα τα οποία έχουν λάβει ε, ελαττωματικό περιεχόμενο ή έχουν πρόβλημα με τον ε, πάροχο της υπηρεσίας. Τώρα για τα υπόλοιπα αγαθά... Ε, έχουμε για παράδειγμα τις πωλήσει ε, εξ αποστάσεως, τις πωλήσει offline και εδώ μιλάμε για το 90% όλων των αγαθών το 90% όλων των αγαθών ε, για τα οποία γίνονται τέτοιου είδους συναλλαγές είναι ακριβώς εμπορεύματα. Άρα λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, έχουμε, έχουμε κάποιες ανησυχίες για τα υλικά αυτά αγαθά. και ίσως οι κανόνες οι οποίοι θα θεσπιστούν θα ε, ισχύσουν μόνο για τις συναλλαγές online. Τώρα για την καταλληλότητα και τον έλεγχο καταλληλότητας όταν προετοιμάζαμε την οδηγία για τις ψηφιακές συμβάσεις για τα υλικά αγαθά είχαμε δύο επιλογές. Ήταν να εναρμονίσουμε και το τι γίνεται offline και οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μνήμη θεσμική από εμένα είπαν πως έγιναν αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν εναρμονιστούν εκεί οι κανόνες και δεδομένου του ότι προετοιμάζαμε την οδηγία στα πλαίσια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και της σχετικής στρατηγικής ήθελα να παρουσιάσω καταρχήν τους κανόνες για τα online και μετά να ακολουθήσουμε με τον έλεγχο καταλληλότητας ε, για να δούμε εάν υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε κάποιο είδους εναρμόνιση και για τις offline πωλήσει. Τα πρώτα στοιχεία θα φτάσουν στα χέρια μας τον ε, Ιούλιο και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας καταναλωτών που κάνουμε τον πρώτο έλεγχο καταλληλότητας δοκιμάζουμε έξι διαφορετικές οδηγίες. Είναι οι πωλήσει B2C οι αθέμπτες εμπορικές πρακτικές, οι εγγυήσει και οι προϋποθέσεις και συνθήκες ε, πώληση είναι οι οδηγίες αυτές. Επίσης η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή που εγκρίθηκε πέρυσι και επίσης από την ψηφιακή εποχή προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω μας ό,τι έχει να παρχαιωμένο, δεν λειτουργεί, πια δεν χρειάζεται και να εστιάσουμε τώρα στα σημεία τα οποία εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν και να ονειρμανίσουμε και τους κανόνες για τις πωλήσει offline. Αυτό το ξεκαθάρισα και στον εισηγητή την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και θα τον ενημερώσω και δεν πρόκειται να του αποκρύψω οποιασδήποτε πληροφορίες που θα προκύψουν στον έλεγχο καταλληλότητας. Ήταν κάπως διακινδυνευμένο από πλευρά μου γιατί δεν ήθελα εγώ να υποσκάψω την όλη διαδικασία α, για τις α, ε, ψηφιακές συμβάσεις για τελικά αγαθά αλλά ήθελα να είμαστε σίγουροι πως κάτι κάνουμε και στην περίπτωση των πωλήσεων offline. Όταν δούμε τη διαφορά μεταξύ off και online, διαδικτυακός δηλαδή και μη, Βλέπετε πως μπαίνουμε σε θέματα καταναλωτικού δικαίου και εκεί το βασικό μας καθήκον είναι ε, να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους σε αυτή τη σχέση. Και τα άτομα που αγοράζουν προϊόντα online είναι πιο τροτά από τα άτομα που πηγαίνουν σε ένα μαγαζί και μπορούν να ψαχουλεύσουν και να ψάψουν τα εμπορεύματα που τους ενδιαφέρουν. Γι' αυτό θέλουμε να καταλήξουμε και σε κάποιους ε, κανόνες αργότερα όμως για τα offline. Αναγνωρίζω βέβαια πως όλο και περισσότερο περνάμε σε μια εποχή ε, μεικτών πωλήσεων offline και online. Δηλαδή πάρα πολλά καταστήματα προτείνουν και online πωλήσει και το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει, για τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας, θα σας τα πω ε, σε διάφορες χρονικές στιγμές. Έχουμε δύο οδηγίες τώρα τον Ιούνιο και μετά έχουμε και τις τέσσερις υπόλοιπες συν ε, αυτή για την οδηγία για τους καταναλωτές και την προστασία τους μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και εκεί θα ήθελα να δω αν χρειάζεται απλούστευση αυτής της νομοθεσίας και ενδεχομένως αντί να έχουμε έξι οδηγίες θα μπορούσαμε να έχουμε μία ή δύο και να καλύπτουμε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους καταναλωτές. Να δούμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία κάπως μπορούμε να την κατευθύνουμε για την εξωτερική διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ που με ευχαριστήσατε, που συγκεντρωθήκαμε και στο θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Ουκρανία, γιατί αυτά είναι ζωτική σημασία για τους Ευρωπαίους. Το σύστημα του δικαστικού για παράδειγμα, και η μεταρρύθμιση σε αυτές τις χώρες της γειτονίας, για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τις χώρες ένταξης είναι πολύ ουσιαστικό για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρικέ σχέσεις. Για την Ουκρανία νομίζω θα τα πούμε αύριο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί ήμουν πολύ πρόσφατα στην Ουκρανία και θα ξαναπάω για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στην Ουκρανία και για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις με τον κατάλληλο και επιτυχημένο τρόπο έτσι ώστε να διώκονται όσοι χρειάζεται. Και πρέπει να σου πω πως θαυμάζω το τι κάνουν όσοι εκεί προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τελειώνει και με ένα μακροπρόθεσμο έργο το οποίο είχε σκοπό να βοηθήσει την Ουκρανία να ε, εισάγει κάποια μέτρα και διατάξεις και ίσως θα μπορούσα από εσάς να εμπνευστώ. Να δούμε δηλαδή τι θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ως νέο έργο και τι τους χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να έχουμε το να στέλνουμε εμπειρογνώμονες στην Ουκρανία και να κάνουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο θα ήταν για μας πολύ καλοδεχούμενο. Θα τα πούμε αύριο. Για την αφηρηγιότητα και τις χρεοκοπίες άκουσα κάποιες ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή ε, μας απασχολεί το θέμα περισσότερο σε εταιρικό επίπεδο. Το 2014 άλλωστε εκδώσαμε τις συστάσεις που καλούν τα κράτη-μέλη να αλλάξουν ε, τις διατάξεις περί αφαιρεγγιότητας και χρεοκοπίας, να δώσουν μια ευκαιρία στους καλούς επιχειρηματίες, να μην στιγματίζονται, να τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, να μπορούν να ξεπεράσουν τις ε, δυσκολίες τους, να γίνεται μια ε, πρώτη αναδιάστρωση πριν φτάσει η εταιρεία σε κρίση, να λαμβάνονται μέτρα. Σύμφωνα βέβαια πάντα με την εθνική νομοθεσία τώρα πρέπει να σας πω πως είναι πραγματικά φρικτός ο αριθμός. 600 επιχειρήσεις την ημέρα κλείνουν. Και στιγματίζουμε την αποτυχία στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω πως αυτοί που πέφτουν δύσκολα ξαναστέκονται στα πόδια τους. Οπότε στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσους έχουν οικονομικές δυσκολίες να συνεχίσουν και αυτά γίνονται στα πλαίσια της ε, ενωσιακής στρατηγικής για τις κεφαλαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, μας απασχολούν οι εταιρικέ χρεοκοπίες αλλά ίσως μπορούμε να δούμε και ε, το θέμα για τα νοικοκυριά, για την ιδιωτική δηλαδή, για την χρεοκοπία ιδιωτών, με συγχωρείτε, και θέλουμε να δούμε τι θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε. Υπάρχει κάποιο νομοθετική πρόταση που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε. Δεν νομίζω πως αυτό θα ήταν σωστό. Είμαι περισσότερο υπέρ του να επενδύσουμε σε καλύτερη γνώση και καλύτερη κατανόηση των οικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνουν ε, τα μεμονωμένα άτομα που δανείζονται από ε, εξωτραπεζικούς θεσμούς και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλες εκστρατείες στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και αυτό. Εγώ ψάχνω την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και το πρόβλημα αυτό είναι το ίδιο για όλους. Δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μην το αντιμετωπίζει. Χρεώνονται σε όλα τα κράτη-μέλη, όλοι, ε, με δυσβάσταχτα δάνεια και είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Οι υπολογισμοί μου είναι πως για το θέμα αυτό της αφηρεγγιότητας και για τις επιχειρήσεις η πρωτοβουλία ε, της νομοθετικής πρότασης θα καταφτάσει στα τέλη της χρονιάς. Ο κύριος φως δεν με χαροποίησε. Ήταν βέβαια οραματικές οι δηλώσεις σας, οι νέες τάσεις, εταιρικό δίκαιο, ψηφιοποίηση, ε, επιχειρηματικός κόσμος κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο. Και το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω τώρα είναι πως είμαστε βέβαιοι πως θέλουμε να βοηθήσουμε τις ε, εταιρείε να είναι πιο έτοιμες για την ψηφιακή εποχή και να εξετάσουμε τις δυνατότητες εισαγωγής πιο συγκεκριμένων εργαλείων που να έχουν στη διάθεσή τους επιχείρηση με ψηφιακό τρόπο λοιπόν να το χρησιμοποιούν και για την ελεύθερη κυκλοφορία και για τη συνοριακή ε, κυκλοφορία στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεργαστείτε μαζί μας εντατικά. Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένη πρόταση για την ε, ε, ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου το φθινόπωρο. Και αυτό με οδηγεί στο να απαντήσω ε, την, την ερώτηση της κυρίας Ρέγνερ για το ΣΟΥΠ, για αυτή την, το είδος εταιρεία. Εδώ θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Και δεν πρόκειται να την αποσύρουμε τη σχετική πρόταση. Εγώ εργάστηκα πάρα πολύ σκληρά για να διαλύσω όλες τις αμφιβολίες για το ποιες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και βεβαίως είμαι ανοιχτή στο να το συζητήσω και με τα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, πιο πολλά χέγγια έτσι ώστε να μην αποτελεί απλή επιχείρηση θηρίδα ή εν πάση μια διαδικασία την οποία θα χρησιμοποιούν καταχρηστικά άτιμοι επιχειρηματίε. Αλλά δεν πρόκειται να αποσύρουμε την πρότασή μας ακόμα. Θέλω πάντως το θέμα του εταιρικού δικαίου και την ψηφιοποίηση να τα θεωρήσουμε μια ευκαιρία για να εξορθολογήσουμε ε, κατάσταση και να βοηθήσουμε τις εταιρείες στο δεύτερο εξάμεινο της φετινής χρονιάς. Τώρα, ε, η διοκτησία και η προστασία δεδομένων είναι το αστικό δίκαιο. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οποιαδήποτε φορά αγγίξουμε κάτι στο αστικό, ξυπνάνε τα κράτη-μέλη. <clears throat> Σίγουρα λοιπόν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, αλλά Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει υποψίες για το ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο είδους ευρωπαϊκό αστικό κώδικα, γιατί δεν είναι κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Κάθε χρόνο θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όπω ξέρουμε έχουμε το στόχο του 40% για τις γυναίκε στα συμβούλια των εταιριών. Έχουμε μπλοκάρει στο Συμβούλιο γιατί υπάρχουν χώρες όπου ήδη υπάρχει αυτή η νομοθεσία όπως η Γερμανία, η Σουηδία και κάποιοι άλλοι που δεν επιθυμούν να μας βοηθήσουν και πολύ για να εγκρίνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτά τα θέματα. Το δικό μου επιχείρημα είναι πάντα το ίδιο. Παρακαλώ πάρα πολύ από τη στιγμή που εσείς είστε προστατευμένοι, βοηθήστε και τους υπολείπους. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την ε, μειοψηφία που μπλοκάρει. Φαντάζεστε ποιοι είναι, έχω ήδη διαβάσει δύο από τους τρεις. Πάντως ελπίζω θα έχουμε εντατικές επαφές και με τις ίδιες εταιρείε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχω πολύ καλή ανταπόκριση από τις εταιρείε, ιδιαίτερα από αυτές που έχουν Αμερικανούς ιδιοκτήτες γιατί έχουν εσωτερικές στρατηγικές ώστε να καλούν περισσότερες γυναίκες όχι μόνο για το, το Εποπτικό Συμβούλιο αλλά και για τα Διοικητικά Συμβούλια γιατί ξέρετε αυτοί μετράνε κέρδη και υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι το μέτρο αυτό της ανάμεξης ανδρών γυναικών νέων και πιο ηλικιαμένων ε, υπάρχουν πλέον αποδείξει ότι όλα αυτά οδηγούν σε περισσότερα κέρδη. Κλείνοντας, υπόσχομαι ότι τις ε, ερωτήσεις που δεν απάντησα θα σας στείλω απαντήσεις γραπτός. Για τους ευάλωτους ε, ενήλικες, γιατί δεν εγκαταλείπουμε την ιδέα. Όχι. Θα είμαι πολύ σύντομη πάντως. Όχι, δεν θα καταλήψουμε. Θα ε, κάνουμε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων. Μεταφράζουμε το κείμενο της Σύμβασης προς τα όλα τα κράτη-μέλη ώστε να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν ακριβώς περί Πρόκειται αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είναι περισσότερο πρόβλημα επικοινωνίας και είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε. Πάντως, ε, ε, για τους υπόλοιπους θα σας δώσω απαντήσεις. Κάτι ακόμα που δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, όπως είπα στον κύριο Βος, γιατί ακόμα γίνεται ε, συζήτηση για το ενοχικό δίκαιο. Μπράσελς 2α. Ναι, θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των παιδιών, ε, να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για αμοιβαία ε, αναγνώριση των αποφάσεων, για την επιτάχυνση της διαδικασίας, για μεγαλύτερη συμμετοχή ειδικευμένων ε, οργανισμών και φορέων, αλλά και για να δημιουργήσουμε σαφείς κανόνες για τον καθαρισμό των δικαστηρίων αλλά και για τους κανόνες για την ε, υιοθεσία. Και θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στις θετές οικογένειες αλλά και, στις, και, και στα ιδρύματα φροντίδας. Να λύσουμε και το πρόβλημα των παιδιών γιατί πολλές που μένουν ε, στα ιδρύματα και τις ακροάσεις των παιδιών ε, Κάποια, θέματα δεν χρονίζουν επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ακροματικές διαδικασίες, ε, τρενάρουν, χρονίζουν. Πολλές φορές είναι οικογενειακές τραγωδίες που δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον του παιδιού και γι' αυτό θέλω να εστιάσω σε αυτά τα ζητήματα στο κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Νομίζω τέλη Ιουνίου ή αρχές ε, Ιουλίου θα είναι έτοιμες οι προτάσεις, θα τις υποβάλω. Τα κράτη-μέλη καλωσορίζουν αυτή την πρωτοβουλία και επίσης ενημερωτικά να σας πω ότι σε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού εστιάζουμε στην γονικές προϋποθέσεις και όχι σε θέματα γάμου. Γιατί ΣΕΤΑ δεν είναι δικό μου θέμα. Λυπούμε. Μπορώ να σας δώσω γραπτή απάντηση, αν δεν έχετε πρόβλημα. Διότι βεβαίως έχω κάποιες πληροφορίες. Και δεν θέλω να σας παραπλανήσω. Μία σύντομη παρατηρήση από την κυρία Χάουτα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίτροπε. Όταν θα κοιτάξετε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για την ανοιχτή αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση, θα δείτε ότι ευτυχώ το θέμα αρμοδιότητα και νομική βάση. Η νομική βάση είναι το άρθρο 98 τη Εθήκης Λισαβόνα. Και έχουμε κατά νου ακριβώ το πώ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η ανοιχτή αποτελεσματική διοίκηση. Και για να σας ε, διαβεβαίωσω. Πρόκειται για ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτά μόνο υπάγονται, αλλά υπάρχουν πάρα, πολλά. Αν ε, σκεφτούμε ότι υπάρχουν και εξωτερικέ υπηρεσίε 48 στον αριθμό. Άρα είναι σημαντικό να με Κοιτάξτε, αυτό είναι αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου κ. Τίμερμαν. Θα το τα μεταφέρω και θα του πω και αυτά που σα είπα εδώ. Ότι με χαρά μου θα βοηθήσω προ την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, έτσι εξαντήσαμε, λέει ο Πρόεδρος, ε, το γύρο των έρωτων απαντήσεων. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή που ήταν μαζί μας σήμερα και προσβλέπουμε και στην αυριανή ακρόαση που και πάλι θα παραστείτε εδώ. So, σας καλωσορίσω και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Μιλάμε για την παρουσίαση της ανάλυσης σε ό,τι αφορά τι δυσυνοριακέ αιτήσει επιστροφή έργων τέχνη που λιαντήθηκαν σε ένοπλε συγκρούσει και πολέμου και λύσει εναλλακτική τη προσφυγή στο δικαστήριο. Ähm, vorstellen wird die eingehende Analyse nun äh, Professor Mark ο καθηγητή Μάρκ Αντζέ από το Πανεπιστήμιο τη Γενέβη θα μα παρουσιάσει την έκθεση αυτή, την ε, εντελεχή αυτή ανάλυση. Έχετε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σα ενδιαφέρεται για το πάρα πολύ επίκαιρο αυτό ζήτημα. Καταρχά, λοιπόν σα ευχαριστήσω που μου αναθέσατε την ανάλυση αυτή και μου δίνετε και την ευκαιρία να σας την παρουσιάσω εν συντομία και φυσικά να την συζητήσουμε και περαιτέρω. Εξ όσων άκουσα, είναι διάφορα τα θέματα που σας απασχολούν στην Επιτροπή σας και έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένω να πρόκειται για ένα επιπρόσθετο ζήτημα το οποίο στο μέλλον θα σας απασχολήσει. The starting point is, um... Το σημείο εκκίνησης είναι η λαιλάτιση ε, έργων τέχνης κατά τη διάρκεια ενοπλών σειράξεων. Αυτό προφανώς ε, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο με μακρά ιστορία και προφανώς ε, έχουμε απευθείας κατά νου τα όσα συνέβησαν στον Δεύτερο Πόλεμο και την εκτενή λαϊλάτηση που έλαβε χώρα τότε. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε και αυτό αποτελεί άλλωστε και έναν από τους στόχους της ανάλυσης αυτής, ότι πρόκειται για ένα θέμα με πολύ, ευρύτερη, πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογή από ότι ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ασφαλώ και αποτελεί ένα πολύ οδυνηρό κεφάλαιο. Αλλά θα θέλαμε να εξηγήσουμε και πιο πρόσφατα περιστατικά. Τέτοιε περιπτώσει λαϊλάτιση ε, στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ιεμένη. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω, μιας και η έκθεσή μου έχει να κάνει κυρίως με τις ε, λαιλατήσεις ένοπλες συγκρούσεις, ασχολείται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και με τις σημερινές συζητήσεις και τις σημερινές ένοπλες συγκρούσεις μάλιστα. Εισαγωγικά, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια προκαταρτικά. Όταν εξετάζουμε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα όπως αυτό, όπως το διαβάσετε και στην έκθεση. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ε, απλούστευσης, όπως ήθιστε σε περιπτώσεις συγκριτικού δικαίου. Ε, κάνουμε κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει επίσης πολλά παραδείγματα. Δεν θα σας τα παρουσιάσω εδώ γιατί θα μακρηγορήσω ιδάλλως, αλλά αν θέλετε μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων Artemis, μία από τις βάσεις δεδομένων που α, χρησιμοποιώ στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Η βάση αυτή Artemis περιλαμβάνει πολλές υποθέσεις λαιλάτισης και αποκατάστασης τέχνης και πολιτισμικής κληρονομιάς και εξετάζει τους διάφορους τρόπους απάντησης των ερωτημάτων αυτών και των ζητημάτων αυτών. Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στο ψητό της έκθεσης. Καταρχά, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, εξέτασα τις νομικές βάσεις για τις ε, αξιώσεις αποκατάστασης και επιστροφής τέχνης και πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι νομικές υποθέσεις είναι πολύ ποικιλές, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά από πλευρά διεθνού δικαίου θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει ό,τι χρειαζόμαστε. Υπάρχουν συγκεκριμένε διεθνεί συμβάσει τη UNESCO, τη UNITRAD, του Συμβουλίου του, τη Ευρώπη που έχει και αυτό επικυρώσει κάποιε σχετικέ διεθνεί συμβάσει. Δεν χρειάζεται να προσταθεί ένα νέο επίπεδο νομικών κειμένων. Ωστόσο, πολύ πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε την εφαρμογή και υλοποίηση των κειμένων αυτών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποίησα κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα στην έκθεση για κάποια συγκεκριμένα εθνικά νομοθετήματα, τα οποία θα ήταν ενδιαφέρον να τα εξετάσουμε αναφέρω δύο. Ένα νόμο των κατοχωρών και ένα νόμο της Ελβετίας της χώρας μου. Τα αναφέρω αυτά ενδεικτικά. Και γιατί είναι τόσο ενδιαφέροντα τα παραδείγματα αυτά, γιατί καταδεικνύουν ότι οι συμβάσει, οι συνθήκε που υπάρχουν και τι οποίε έχουν επικυρώσει πιο πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Οι συνθήκε λοιπόν αυτέ ε, υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίησή του, στην εφαρμογή του. Εφόσον έχουν υλοποιηθεί, τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά. Το παράδειγμα των κάτω χωρών καταδεικνύει ότι υπάρχει μια σχετική νομοθεσία. για την εφαρμογή του πρώτου πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης του 1954, που πραγματεύεται την προστασία της τέχνης και της πολιτισμικής κληρονομιάς σε περίοδους πολέμου και το πρωτόκολλο πραγματεύεται το παράνομο εμπόριο που ακολουθεί συνήθως μετά από την κατοχή μιας χώρας ε, για τη σημερινή εποχή, για παράδειγμα στο Ιράκ, στη Συρία. Καμία από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη αυτή δεν έχουν εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Χάγης, εκτός από τις κάτω χώρες, οι, οποίοι, οι οποίες και το 2007 ενέκριναν μια νομοθεσία που εγκρίνει το πρωτοκόλλο αυτό, που ε, υλοποιεί το πρωτοκόλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πρωτόκολλο λοιπόν του 54 υλοποιήθηκε από μία μόνο χώρα και τι λέει λοιπόν, ότι οι κανόνες του πρωτοκόλλου είναι άμεσα εφαρμόσιμοι. Ε, πρώτο λοιπόν ε, παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα στην Ελβετία. Προσφάτως ανεκρίθηκε μια νομοθεσία για την ε, ύπαρξη ασφαλών λιμένων σε περίπτωση ενόπλων σειράξεων. Αυτό είναι γνωστό σε διεθνέ επίπεδο. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό και στην Ένωση Διεθνού Δικαίου και σήμερα λοιπόν το Safe Havens έχει εγκριθεί ω νομοθεσία στην Ελβετία, προωθείται και στην Γαλλία. Σε περιπτώσεις όπου τα έργα τέχνης λοιπόν μπορούν να προστατευθούν σε περιπτώσεις ενόπλων σειράξεων, σε ουδέτερα μέρη, σύμφωνα με τη διεθνή συμβάσεις, σε, σε ό,τι αφορά ε, εργατέχνη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια από την UNESCO. Και εκεί λοιπόν μπορούν να φυλάσσονται τα εργατέχνη υπό προστασία. Ενδιαφέρουσα λοιπόν και αυτή η νομοθεσία και ενδεχομένως να θέλετε και εσείς ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλογιστείτε μια τέτοια λύση, η οποία ενδεχομένω να είναι απαραίτητη. Σε ό,τι αφορά το soft law, το ήπιο το δίκαιο, θα είμαι σύντομο. Δεν πραγματευόμαστε μόνο την εθνική νομοθεσία και οι, Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Δεν χρειάζεται να σα μιλήσω για αυτού. Του γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμένα. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το, τα στοιχεία του soft law περιλαμβάνονται σαφώς στον τομέα αυτό. Το 1998, το 1998 έγινε μια συνάντηση των πολιτιών στην Ουάνσιγκτον, όπου και εγκρίθηκαν οι αρχές της Ουάσιγκτον για τα έργα τέχνης που είχαν κατάσχει οι Ναζί. Οι αρχές λοιπόν αυτές τι προσπαθούν να κάνουν, να διευκολύνουν την διαδικασία επιστροφής τέχνης που είχαν λαιλατηθεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αρχές λοιπόν αυτές ε, αναπτύχθηκαν περαιτέρω και στην Πράγα μεταξύ άλλων το 2009 εγκρίθηκε και μια σχετική διακήρυξη. Βάσει λοιπόν των αρχών αυτών διάφορες ε, χώρες έχουν εγκρίνει διάφορες συγκεκριμένες διατάξεις που διευκολύνουν και δίνουν τη δυνατότητα για την αποκατάσταση και την επιστροφή τέτοιων εργοτέχνης που λέει λατήθηκαν, κατασχέθηκαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη λοιπόν και αυτή από πλευρά ε, soft law, ήπιου δικαίου. Θα συνεχίσω γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και δεν θέλω να σα απασχολήσω πάρα πολύ. Να κοιτάξουμε ποιε είναι οι νομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο κόσμο. που έχει πέσει θύμα τέτοια λαϊλάτηση τέχνη. Είτε είναι ιδιώτε, είτε είναι κράτη. Μέσω, για παράδειγμα, παράνομων αρχαιολογικών ανασκαφών. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Καταρχάς, η ιδέα, η έννοια της τέχνης, ε, λέει, λατημένης τέχνης, θα πρέπει να οριστεί. Δεν είναι απλό να οριστεί. Είναι και πολύ πολύ σύνθετος ο ορισμός του τι είναι καταναγκαστική α, αγοραπολισία. Γιατί ουσιαστικά το αποτέλεσμα το ίδιο είναι και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση της λαϊλασίας και στην περίπτωση της καταναγκαστικής ε, ε, πώληση. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει μια μέθοδος αποκατάστασης. Δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς των περιορισμών γιατί φυσικά ο χρόνος περνάει, μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για πράγματα που έχουν συμβεί πριν από πολύ καιρό, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και πιο πριν σε κάποιες περιπτώσεις και συχνά όταν οι, τα έργα τέχνης κυκλοφορούν, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί και αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο το οποίο συχνά αντιμετωπίζουν τα θύματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, σήμερα συζητούν ένα ομοσπονδιακό κάθεστος. Σα το έχω βάλει και στο παράρτημα. Είναι το προσάρτημα υπερθυμών 4. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί στην γεωρουσία των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2016 προκειμένου να υπάρχει στι ΗΠΑ ένα ενιαίο σύστημα για την περίοδο περιορισμού για την υποβολή αξιώσεων για τέτοια έργα τέχνης που έχουν λαϊλατηθεί. Και άρα προτείνεται μια ε, περίοδος έξι ετών για την υποβολή της αξίωσης αυτής από τη στιγμή που ανακαλύπτεται το που βρίσκεται το έργο τέχνης και εντοπίζεται. Άρα το θύμα έχει έξι χρόνια στη διάθεσή του. Και είναι ενδιαφέρον τώρα ότι υπάρχουν διάφορες πολιτείες οι οποίες προσπαθούν να επεκτείνουν αυτή την περίοδο την εκθέτηση των εξήτων. Για ότι, σε ό,τι αφορά τα θύματα και τους απογόνους των ε, θύματων, σε ό,τι αφορά τα περιπτώσεις σύγκρουσης ε, νομοθεσίας και ε, προβλημάτων δικαιοδοσίας. Προφανώς αυτά κυκλοφορούν ως εργατέχνης και το πιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο είναι ένα θέμα, καθώς και το εφαρμόσιμο δίκαιο. Μιλάμε για θέματα ιδιοκτησίας κυρίως. Η αρχή είναι το lex reisite. Ισχύει το δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται το αντικείμενο. Αυτός ο κανόνας όμως μπορεί να έχει συχνά αρνητική επίπτωση για αυτούς που ζητούν αποκατάσταση. Γιατί ο νόμος ε, του τόπου όπου έλαβε χώρα η συναλλαγή, η επιστροφή, ή μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι ευνοϊκός, γιατί μπορεί να προστατεύσει την καλή πίστη του αγοραστή. Μια αρχή που ισχύει σε, πολλά χώρα, πολλές χώρες. Άρα κάποιοι ζητούν ενδεχόμενη ανατροπή του λέξε ρέισίτε για να περάσουμε στο λέξη Origine, δηλαδή στην νομοθεσία της χώρας προέλευσης, η οποία και ισχύει πιο πολύ για αρχαιολογικά ευρήματα, σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, παράνομων ανασκαφών. και ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να ισχύει, πιο πολύ το δίκαιο της προέλευσης. Τελευταίο εμπόδιο και από ιδεολογικής άποψης για πολλούς είναι το θέμα της καλής πίστης. Συχνά ξέρετε. Ενδεχομένως ο ακούραστης να έχετε με καλή πίστη να κάνετε συναλλαγή. Ποια είναι λοιπόν τα συμφέροντα θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του αγοραστή καλή πίστη. Η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία το προστατεύουν αυτό ως αρχή ή προτιμούμε να προστατεύσουμε την αξίωση του ατόμου το οποίο έχει στερηθεί ή του απογόνου του. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ βασικό και πολύ δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το ζήτημα αυτό το έχετε πραγματευτεί και εσείς εδώ. Και υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχει και μια οδηγία του 2014 για την επιστροφή νόμος διακινούμενων αντικειμένων. Ιδέως επιμέλεια ορίζεται στο άρθρο 4 της σχετικής οδηγίας. Για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, η προέλευση. Η προέλευση είναι βασικό ζήτημα εδώ. Όταν έχει κλαπεί, έχει εξαφανιστεί ένα έργο τέχνης και επανεμφανίζεται πολλά χρόνια μετά. Ε, εδώ λοιπόν τύφλει το θέμα αυτό. Τα κράτη, τα μουσεία, οι εξειδικευμένε οργανώσεις, οι έμποροι, όλοι έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα της προέλευσης. Από πού προήλθε αυτό το έργο τέχνης και πώς μεταφέρθηκε από τον ενδιακτήτη σε άλλον. Θέματα έρευνα για την προέλευση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα σε διάφορα κράτη. Ακριβώς για το ζήτημα αυτό προσπαθώντας να βοηθήσουν όσους έχουν τέτοια ζητήματα. Για να εντοπιστεί λοιπόν η προέλευση τέτοιων εργών τέχνης και για να αποτρέπονται οι κλοπές. Η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ιδιαίτερα προγράμματα σε ό,τι αφορά την προέλευση έργων τέχνης. Ασφαλώς η δυσκολία έγκυται στο ότι και αυτή η έρευνα έχει κάποια όρια και επίσης η χρηματοδότηση της έρευνας αυτής δεν επαρκεί πάντα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα διαφωνιών, πώς επιλύονται. Ως ε, ως ε, δικηγόρος ασφαλώς ε, θα αναφέρω και τις δικαστικές αγωγές. Ε, Βεντιλή vs. Giuseppe, ό,τι αφορά το Λούβρο στη Γαλλία, όπου η απόγονη μιας οικογένειας που είχε πέσει θύμα λαϊλασία έργων τέχνης, στη δεκαετία του 40, κατάφεραν να πετύχουν την επιστροφή των έργων τέχνης τους πήρε όμως πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τους κόστησε και πάρα πολλά χρήματα και ήταν δύσκολη η υπόθεση. Πολλοί λοιπόν διατείνονται ότι θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικέ μέθοδους ε, επίλυσης των διαφωνιών. Θα πρέπει να μπορούμε να καταλήγουμε σε κάποιες λύσεις και πέρα από τα δικαστικά, από το δικαστική οδό. Εγώ εξέτασα διάφορους τέτοιους τρόπους, διατησία, συμφιλίωση, διαπραγμάτευση και διατησία. Στην διατησία πρέπει να πω ότι δεν βλέπουμε τέτοιε πολλέ περιπτώσει στον τομέα αυτό. Ενδιαφέρον, γιατί κατά πάσα πιθανότητα όταν ανακύπτουν αυτέ οι υποθέσει, δεν υπάρχει κάποια ρήτρα διατησία, δεν υπάρχει κάποια σχετική σύμβαση και άρα είναι δύσκολο να καταλέξουν σε κάποια συμφωνία τα μέρη. Σε κάποια συμφωνία διατησία, δηλαδή. Αλλά η διαβούλευση, η συμφιλίωση και η διαπραγμάτευση ε, χρησιμοποιούνται. Και αυτό το επιβεβαιώνει και η βάση δεδομένων Artemis. Κάποιες διεθνείς οργανώσεις έχουν επιδείξει ενδιαφέρον σε θέματα διαμεσολάβησης στο συγκεκριμένο θέμα, η WIPOL, η Παγκοσμία Οργάνωση για την Πνευματική διακτησία, πρότεινε πλέον συγκεκριμένες διατάξεις για θέματα διαμεσολάβησης σε συνεργασία με την ICOM, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Είναι κάτι μάλλον καινούριο λοιπόν αυτό ως πρόταση. Γιατί λοιπόν οι μηχανισμοί αυτοί είναι τόσο ενδιαφέροντες. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω γιατί εξειδικαστική επίλυση είναι ενδιαφέρουσα λύση. Αυτό που είναι όμως ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι βρίσκονται πολύ πρωτότυπες λύσεις και από τη δικασία διαμεσολάβησης και από τη διαδικασία ε, διαπραγμάτευσης και συμφιλίωσης. Και τι εννοώ. Δίκαιες λοιπόν λύσεις. Δίκαιες λύσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό προωθούν και οι αρχές της ε, Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Δίκαιη λύση και σωστή λύση. Και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ε, προϋποθέτει και ένα ανοιχτό χαρακτήρα, μια κάποια ευελεξία αντιμετώπισης και προσέγγισης της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα θύματα. Αυτές λοιπόν οι λύσεις, οι σωστές και δίκαιες λύσεις εγκρίθηκαν και προωθήθηκαν και επιτεύχθηκαν σε διάφορες περιστάσεις από τους υπεύθυνους διαβούλευσης, συμφιλίωσης και διαπραγματεύσεις. Υπάρχει αφενός ε, η λύση της αποζημίωσης. Αλλά και το θέμα της ε, συνδιοκτησίας, στην σελίδα 4 το βλέπετε αυτό. Παραδείγματα για το πώς επιλύονται δύσκολες περιπτώσεις μέσω συνδιοκτησίας. Εδώ έχω κάνει μεγάλη έρευνα, πρέπει να σας πω. Και για να περάσω στον κλάδο σύσταση ε, πολιτικών, στον, στην ενότητα αυτή. Τρεις προτάσεις έχω να κάνω εδώ. Καταρχά. η επιδίωξη μιας ε, ενιαίας μορφής των λύσεων, μιας καθολικής μορφής λύσεων, μέσω ε, ενιαίων ομοιογενών κανόνων σε διεθνές επίπεδο για την επίλυση των διαφωνιών. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα προκειμένου όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ένα κοινό κώδικα για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων. Αυτό νομίζω ότι θα αποτελούσε με ένα πρώτο βήμα για την ομοιογένεια και θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει το Lex Originis, όπως είπα και προηγουμένως. Δεύτερο στοιχείο, δεύτερη σύσταση την οποία θα ήθελα να κάνω. Να επιδιώξουμε ομοιόμορφα πρότυπα στην Ένωση. Αυτό είναι θέμα ουσιαστικού δικαίου, θέμα δεούσης επιμέλειας, για παράδειγμα. Ορισμού όλων των στοιχείων αυτών. Και προτείνω στην έκθεση να ληφθούν κάποια μέτρα στα κράτη-μέλη για να επικυρωθούν τα ήδη υφιστάμενα νομοθετήματα, ήδη υφιστάμενες συνθήκες, όπως για παράδειγμα το safe havens ε, που ανέφερα και προηγουμένω, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη θα αντιληφθούν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα τι συμβάσει τι οποίε έχουν προσυπογράψει, ακολουθώντα τα παράδειγμα των χωρών. Σε ό,τι αφορά τις αξιώσεις και τις δικαστικές καταγγελίες και αγωγές, και σε δικαστηρία αλλά και σε άλλες ε, οργανώσεις. Θα έλεγα να, να εγκριθούν ενιαία πρότυπα θεούσης επιμέλειας υπό την έννοια του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2014 και επιπροσθέτως ενδεχομένω ε, ένα συγκεκριμένο κώδικας για τους περιορισμούς, όπως εγκρίθηκαν και από τις είπα, από σας είπα προηγουμένως. Τέλος. Ένα διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο ενδεχομένω δεν ενδιαφέρει να λεφτεί υπόψη. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε να συσταθεί μια ειδική πλατφόρμα, ένα ειδικό σώμα που θα μπορούσε να πραγματευτεί ακριβώς το δύσκολο αυτό ζήτημα της ε, τέχνης, των έργων τέχνης που έχουν κλαπεί πριν από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα τέτοιο λοιπόν συμβουλευτικό σώμα θα μπορούσε να παρέχει αρρωγή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση διεθνών συμβάσεων. Θα μπορούσε να συνδράμει και στα δικαστήρια και άλλες ενώσεις. Και τέλος, νομίζω ότι θα μπορούσε να επιλύσει διάφορες ε, συγκρούσεις και διαφωνίε βάσει λύσεων διαμεσολάβηση και συμφιλίωση. Άρα, συνοπτικά, νομίζω ότι πολλά μπορεί να γίνουν ακόμα και θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, ένα σημείο καμπή, θα έλεγα, και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να παρέμβω στο θέμα αυτό, στο σημείο αυτό. Και θα Ξέστηνα πραγματικά να ληφθούν μέτρα και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ε, σε περίπτωση που υπάρχουν ε, απορίες σχετικά με την παρουσίασή μου. Ελπίζω να μην μακρηγόρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η παρουσίαση της κατάστασης και θα ήθελα και εγώ προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι σας αφήσαμε να, περιμένουν, να περιμένετε, γιατί η προηγούμενη παρουσίαση πήρε λίγο παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Και έτσι να περάσουμε στι ερωτήσει. Ο κ. Καβαντά. Merci, Président. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς για την έκθεση αυτή και για την πολύ διαφωτιστική προσπάθεια που κάνετε. Η γραμματεία της δικής μας Επιτροπής ήδη μας έχει ενημερώσει πριν από κάποια λεπτά πως το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί το 2003 στο Κοινοβούλιο από τον Βίλι Κλέρκ. Νομίζω ότι εκτός από την οδηγία που ε, ψηφίσαμε γιατί δεν είναι ο κύριος Δεκλέρκ εδώ, εκκρεμεί ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, πάντα καυτό, με απήχηση στην κοινή γνώμη, γιατί πρόσφατα ένας Αμερικάνος παραγωγός έκανε μία πολύ γνωστή ταινία για το θέμα αυτό, The Monuments Man. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, εσείς που είστε ειδικός Η UNESCO είναι η καλύτερη βάσο, βάση με συγχωρείτε, για να γίνεται διαιτησία στα θέματα αυτά. Θεωρείτε πως είναι το κατάλληλο επίπεδο και θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δικάζει να αποφασίζει δηλαδή. Γιατί όταν αποφασίζει κανείς να στήσει ένα δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτό έγινε με τη συμφωνία των ε, κρατών ε, μέσω του ΟΗΕ. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε αυτή τη λαιλασία των ε, πολιτικών αγωθών, ίσως ο ΟΗΕ θα ήταν το κατάλληλο βήμα. Νομικά λοιπόν, εάν προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσατε εσείς να συστήσετε κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως είναι το κατάλληλο βήμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και είτε να εκδικάζει είτε να με αποτελεσματικό τρόπο να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους υποθέσεις όταν πρόκειται για διαιτησία. Ε, Σας ευχαριστώ κύριος Κρίστερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση των προβλημάτων αυτών σε ό,τι αφορά την τα έργα τέχνη και για άλλα τα νομικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Δύο ερωτήσει. Καταρχάς, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη, μάλλον υπάρχει αύξηση των νομικών αυτών υποθέσεων για τέτοια κλαμμένα έργα τέχνη και θα μπορούσατε να μας εντοπίσετε σε ποιον τομέα υπάρχει αυτή η αύξηση ενδεχομένω. Δεύτερη ερώτηση. Μα είπατε ποιε είναι οι συστάσει σα προ του πολιτικούς. Εμείς ως Ευρωπαίοι οι ευρωβουλευτέ. έχετε να μα απευθύνετε κάποια συγκεκριμένη σύσταση ή πιστεύετε ότι στην τελική ανάλυση είναι θέμα του ΟΗΕ και στην τελική ανάλυση πιο αρμόδια είναι ενδεχομένω στο διεθνή όργανα. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και εγώ έχω δει τρει ερωτήσει, επιτρέψτε μου. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σε ένα πλαίσιο πολέμου, αταξίας, ε, καταναγκαστικών συναλλαγών υπάρχουν και διαστάσεις σε ό,τι αφορά την ιστορία. Καταρχάς, υπάρχει κάποια παραγραφή. Αν όχι, θα έπρεπε να προβλέπετε μια ενός είδους παραγραφή σε ό,τι αφορά τα αξιώσεις. Κατά δεύτερον, ακούγοντας τι έγινε στην περίπτωση, στην υπόθεση Google στη Γερμανία. Σας έκανε κάτι εντύπωση στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και μία τρίτη ερώτηση. Είχατε βάλει ένα ερωτηματικό μετά τις διεθνείς πλατφόρμες και τι διεθνείς επιτροπές. Γιατί Θεωρείτε ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο αυτό απόλυτο νομική σκέψη, για κάποιο νομικό δισταγμό. Κύριος Μπερζερόν, παρακαλώ. Η κυρία Μπερζερόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί χρησιμοποίησατε τον όρο πολιτιστικά. Το έργα τέχνης είναι μειωτικό, κατά τη γνώμη μου γιατί καταρχήν είναι υποκειμενική η τέχνη και δεύτερον τι σημαίνει αντικείμενα τέχνης, γλυπτική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική για τη Γαλλία. Άρα λοιπόν το να ελελετήσει κανείς ένα αφρικανικό νεκροταφείο ε, και να αφαιρέσει από εκεί σύμβολα ή να κλέψει αντικείμενα από το Περού δεν θεωρείται ε, ε, πώς έχει κλέψει κανείς εργατέχνης, αλλά πολιτιστικά αγαθά. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε αυτή την αντικατάσταση εδώ, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε έναν ορισμό των ε, όσων αντικειμένων θέλουμε να καλύψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εξαρτήσαμε λοιπόν το κατάλογο των ομιλητών. Σας παρακαλώ να πάρετε και πάλι το λόγο για να απαντήσετε. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Δεν ξέρω ποια είναι η παράδοση εδώ. Πρέπει να απαντάς στις ερωτήσεις στη γλώσσα που έγιναν. Α, είμαι ελεύθερος να επιλέξω. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, μπορώ να απαντήσω στον κύριο Καβαντά στα γαλλικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πού αναφέρεστε στο παρελθόν. Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Και στην ταινία αυτή του George Clooney την οποία πραγματικά θα σας αισθήσω να πάτε να δείτε. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, υπάρχει κι άλλη μια ταινία για την υπόθεση Altman, στην οποία αναφέρομαι στην έκθεση, που είναι η Woman in Gold, η γυναίκα που φοράει χρυσά, που είναι πολύ καλή και παραστατική. Και είναι μια μεγάλη επιτυχία μιας πραγματικά αξιοθαύμαστης γυναίκας θα είναι η UNESCO όντως ο τόπος, ο κατάλληλος για να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους δομή διετησίας. Το πρώτο στοιχείο στην απάντησή μου είναι πως υπάρχει ήδη στα πλαίσια της UNESCO μια διακυβερνητική επιτροπή για την επιστροφή έργων πολιτιστικών, να το πω πολιτιστικών αγαθών. που αφαιρέθηκαν από ή εκλάψαν από κράτος με δικαιοδοσία διαιτητική. Δηλαδή, μπορεί να διαμεσολαβήσει ε, για να λύσει θέματα μεταξύ κρατών για πολύ πολιτικά ζητήματα η UNESCO είναι μια, ένας καταπληκτικός θεσμός, αλλά το να πούμε πως θα έπρεπε η UNESCO να δημιουργήσει μια επιτροπή διαιτησίας ή κάποιο είδους δικαστήριο που θα λύνει αυτές τις ε, διαφορές, δεν είμαι σίγουρος. Και δεν είμαι σίγουρος πως αυτός είναι και ο στόχος τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Σίγουρα δημιουργήσαμε το Διεθνές ε, Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το Διεθνές Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να εκδικάσει και υποθέσεις, για παράδειγμα, πολιστικής γενοκτονίας, και αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτή τη στιγμή η, τρέχει μια διαδικασία στο Διεθνές Αυτό Δικαστήριο, Άρα λοιπόν σχετίζεται με το όσο συζητάμε. Το κατά πόσο θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα διεθνές δικαστήριο που θα δικάζει τέτοιου είδους υποθέσεις δεν είμαι σίγουρος. Ίσως δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Και εδώ θα ασχοληθώ με το τελευταίο ζήτημα που ετέθη, που είναι το ερωτηματικό που έχω βάλει εγώ. Στο τέλος της πρότασής μου, για το κατά πόσο χρειάζεται ένα συμβουλευτικό όργανο, μια διεθνής πλατφόρμα. Νομίζω αυτό θα ήταν πιο εύκολο, μια λιγότερο επίσημη αρχή γιατί ένα δικαστήριο νομίζω ή έστω μια επιτροπή διαιτησία θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο σχέδιο και θα προτιμούσα κάτι πιο ευέλικτο σαν σχήμα. Έτσι ώστε να μην ε, θίξουμε την όλη διαδικασία προσπαθώντας να είμαστε υπερφιλόδοξοι. Α είμαστε πιο μετρημένοι και μην έχουμε ένα ειδικό δικαστήριο για κάθε χώρο που υπάρχει και θέμα που προκύπτει. Ας διατηρηθούμε λοιπόν στα επίπεδα αυτής της ιδέας για μια πλατφόρμα που θα είναι ένας τόπος διαβούλευσης, συμβουλής, αλλά όχι δικαστηρίου. Ο κύριος Κώστερς τώρα μίλησε για την αύξηση των υποθέσεων, ναι. Απαντώ πως ναι. Όντως αυξάνονται. από τα τέλη της δεκαετίας του 90 όπου έχουν ανοίξει τα αρχεία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και με τα θέματα που προέκυψαν κυρίως με την Ελβετία ανακαλύψαμε πως υπάρχουν όλο και περισσότερα έργα τα οποία δεν, έχουν, δεν επιστράφησαν αμέσως μετά τον πόλεμο, όταν έδρασαν οι Monuments Men, είτε αργότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ε, εγκρίθηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο και έχουμε πολλές περιπτώσεις έργων που δεν έχουν επιστραφεί και που θα μπορούσαν να έχουν επιστραφεί. Έχουμε το νομοσχέδιο το αμερικανικό που μιλάει για 650.000. Εντάξει, υπολογισμό είναι. Αλλά είναι ένας αριθμός τον οποίο έχουν, δεν τον έχουν εφεύρει. Οπότε είναι πάρα πολλά, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα, η συγκεκριμένη σύσταση που θα έκανα εγώ προσωπικά για την Ένωση θα ήταν κανόνες για το θέμα της παραγραφής. Εάν θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για το νομικό πλαίσιο εδώ, θα πρέπει οι κανόνες που θα προτείνουμε να είναι σαφείς και κατά τη γνώμη μου το βασικό φρένο που φρενάρει τα θύματα τέτοιου είδους λαιλασίας είναι το θέμα της παραγραφής. Οπότε η δική μου σύσταση είναι να προτείνουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για το ζήτημα αυτό. Και μετά βέβαια υπάρχει και το θεσμικό κομμάτι, όπως είπα και προηγουμένως, ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό, όχι όμως απαραίτητος δικαστήριο. Να περάσω λοιπόν και στην ερώτηση του Προέδρου μιλήσατε για την παραγραφή κι εσείς, έχω την εντύπωση πως το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό προτείνω να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αυτό, να το αντιμετωπίσετε και βέβαια τι γίνεται όταν έχει αποκτήσει κανεί καλή την πίστη κάποιο τέτοιο έργο. Και τι γίνει ε, αν έχει, ε, ε, αν έχει επιδειχθεί η απαραίτητη μέρημνα η απαραίτητη επιμέλεια. Και εδώ θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερη σάρκα και οστά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή όχι μόνο στην παράγραφη, αλλά και στην απαραίτητη φροντίδα ε, στα πλαίσια της αγοράς έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών. Έχουμε την υπόθεση Γκούλιτ που εκτενέστατα αναφέρθηκε στην επικαιρότητα στην ε, Γερμανία και στην Ελβετία, γιατί το Μουσείο της Βέρνης είναι το μουσείο στο οποίο στεγάζεται η συλλογή αυτή ε, του γιου του εμπόρου ε, του, κυρίου Ικλέρ και καταλαβαίνετε πως είναι ένα μάθημα αυτό που μας δίνει η υπόθεση που έχει να κάνει με το κεφάλαιο στο οποίο το προηγουμένως που είναι η προέλευση και το κατά πόσο μπορούμε να ερευνήσουμε την προέλευση και η υπόθεση αυτή αποδεικνύει σε ποιο βαθμό οι έρευνες για την προέλευση κάποιων έργων τέχνης είναι σημαντικές το μουσείο κληρονόμησε τη συλλογή και οι, οργανισμοί αυτοί θα έπρεπε να ψάξουν να δουν αν αυτή η συλλογή ε, που έχει πάνω από 1.400 έργα ε, στεγάζει και κάποια τα οποία αποτελούν αντικείμενο λαιλασίας. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε διευκολύνει την δουλειά όσων αυτή τη στιγμή σήμερα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους συλλογές. Να πω λοιπόν πως υπάρχει ένα ερωτηματικό και να πούμε ότι είναι καλή ιδέα να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που θα ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και για την τελευταία σας ερώτηση κυρία μου, για το τι σημαίνει πολιτιστικά αγαθά και αν θα πρέπει να λέμε εργατέχνης, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Ξεκινήσαμε με τα εργατέχνης γιατί αυτά είχαμε κατά νου, αλλά βεβαίω θα πρέπει να εξετάσουμε και με πιο διευρυμένο τρόπο το θέμα. Ξέρετε τη σύμβαση της UNESCO, τη σχετική, και γνωρίζετε και την ε, οδηγία για την επιστροφή αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωση. όλα τα κείμενα αυτά μιλούν πάντα για πολιτιστικά αγαθά ή για ε, εθνικού θησαυρού. Ας μην περιοριστούμε μόνο στα έργα τέχνης. Και εκεί θα συμφωνήσω και πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια επερώτηση από τον Στάνφο Καβαντά. Συγγνώμη, αλλά όπως και αρκετοί συνάδελφοι δεν, ε, δεν ε, έχω ικανοποιηθεί απόλυτα, οπότε θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και την εμπειρογνωμοσύνη σας. Όλη η ιστορία της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών είναι η προθεσμία παραγραφής. εσείς τι πιστεύετε, ποια θα πρέπει πιστεύετε να είναι η προθέσμια αυτή, δεδομένης της φύσης της κλοπής, της λαιλασίας, ε, δηλαδή και στη διάρκεια πολέμων, τι προθέσμια θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε αποδεχτή. Αν αναφερθώ στα πιο επενδυτικά κράτη όσον αφορά την πνευματική διεκτησία, είναι και 70 χρόνια, ας πούμε για τα, ε, τα απόρριτα αρχεία είναι 50 χρόνια. Ένα αιώνα θα ήταν μια καλή θέση να υπερασπιστεί κανεί. Παραγραφή δηλαδή πέρα από τον έναν αιώνα, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε την υπόθεση. Ένα αιώνα ανάμεσα στην λαϊλασία και την στιγμή τη δικαστική ε, δίωξη. ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά όχι μόνο. Όντω, πιστεύω ότι η έννοια του αιώνα θα ήταν καλή από τη στιγμή της κλοπής. Τίνω να συμφωνήσω με αυτή την ιδέα. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα με το θέμα της προθεσμίας διαγραφής είναι και η στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε πότε ξεκινάει αυτή η προθεσμία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με την Αμερικανική πρόταση είναι ότι θεωρούν την αρχή τη προθεσμία, μάλλον η προθεσμία ξεκινά μόνο και μόνο από τη στιγμή όπου το θύμα ή ο απόγονός του γνωρίζει πού βρίσκεται το ε, ε, πολιτιστικό αγαθό και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να αυτό να γίνει δηλαδή και 100 χρόνια, πολύ περισσότερο από 100 χρόνια μετά. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια μακρά προθεσμία συν συγκεκριμένη προθεσμία για την αρχή της έναρξης της προθεσμίας αυτής. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να το συζητήσουμε περαιτέρω και να σας δώσω όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε για το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και σα σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμα και για την ε, υπομονή σας και για την παρουσίαση αυτού του πολύ, πολύ σύμφετου θέματος. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα μικρό καλούπι και να προβλέψουμε δυνατότητες για δεκαετίες αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 6, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της οδηγιας 2736, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης συνεργού συμμετοχής των μετόχων και της Οδηγίας 2013-34 όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εσωτερικής διακυβέρνησης. Η συζητήση, ο συνάδελφος Κόμφεράτε και μιας και έχει περάσει πολύ η ώρα, χωρίς όμως ε, να θέλουμε να μειώσουμε και την σημασία των επιτευγμάτων σας ε, και τις εργασίες σας, θα θέλω να σας καλέσω σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, να μας παρουσιάσετε τα καθέκαστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι συντομότατος. Εξάλλου, είμαστε σε μια φάση της συζήτησης ε, που μου το επιτρέπει αυτό. Γιατί, όπως θα θυμούνται οι συνάδελφοι, η πρόταση της Κομισιόν χρονολογείται τον Απρίλιο του 2014. Ψηφίσαμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2015 και έκτοτε άρχισαν οι τεχνικές επαφές και στη συνέχεια οι τριμερείς διάλογοι. Ο πρώτος με την Λουξεμβουργική Προεδρία και μετά με την Ολλανδική. Φτάσαμε σε αυτή τη φάση όπου το πρώτο τμήμα της πρότασης του Κοινοβουλίου μετατράπει πρώτα σε τεχνικές συμφωνίες, μετά σε ε, πολιτικές συμφωνίες με το σχέδιο γνωμοδότησης που έχουμε υποβάλει. Έχουμε ιδιορίσει τα όσα αφορούν τον εντοπισμό των μετόχων, τη διευκόλυνση της ψήφου τους, τη διαβίβαση των πληροφοριών, καθώς και τη διαφάνεια του κόστους. Επίσης, συμφωνήσαμε ε, τους κανόνες που αφορούν τους συμβούλους ε, τους proxy advisors. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την Ολλανδική Προεδρία που ήταν διαθέσιμη και έδωσε σημαντική ε, βοήθεια για την αναζήτηση αυτών των ε, συμφωνιών. Βέβαια, αντιμετωπίσαμε και ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχαμε προβλέψει, δηλαδή το πού θα πρέπει να τοποθετηθεί εκείνο το θέμα που αφορά την αναχώρα έκθεση που όπως θα θυμάστε ήταν, μάλλον ερωτήμα που από την Επιτροπή μας στο κείμενο που αφορά την οδηγία για τους μετόχους. Οι κανόνες αναχώρα δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόταση της Κομισιόν ε, τις ανακτήσαμε και τις εγκρινέκρινε και ολομέλεια. Τώρα, στη συζήτηση που έχουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ε, επελήθη το θέμα γιατί η πλειοψηφία των ε, πολιτικών δυνάμεων που αντιπροσωπεύονται σε αυτή την στην Επιτροπή μέσω των σκιωδών θεωρούν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυτοί οι κανόνες στην οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των μετόχων διότι όλα όσα έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και την φορολογική πίστη είναι σημαντικά στοιχεία αξιολόγησης για όποιους θέλουν να επενδύσουν σε μια επιχείρηση και να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Φτάσαμε σε αυτή τη συμβαστική λύση, τη μεθοδολογική συμβαστική λύση. Συνεχίσαμε στην πολιτική και τεχνική σύγκριση για το σύνολο της οδηγίας και για την ώρα αναστήλαμε αυτό το θέμα του χώρου του, της αναχώρας έκθεσης, ώστε να δούμε πώς και πότε θα εξελιχθεί η συζήτηση εκεί όπου επέλεξε η Κομισιόν. Ξέρετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από πλευρά τη Κομισιόν για την τροποποίηση των προηγούμενων κανόνων ακριβώ για το ε, αναχώρα, τις αναχώρα ε, ε, εκθέσεις, αναφορές. Συζητάμε λοιπόν για τα όσα έχουν μείνει σε κρεμότητα που είναι σημαντικά, αλλά είμαι αισιόδοξο γιατί θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Αφορούν τη διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών assets, τα μέτρα για τις ε, συναλλαγές συνδεδεμένων ε, μερών και μετά έχουμε τις κατεξιοδότητες συμπράξεις ε, για τη μελλοντική εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις στους επόμενους μήνες και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε για όλα όσα αφορούν τους μετόχους. Ε, ε, εν τω μεταξύ θα δούμε πού και πώς έχει φτάσει η συζήτηση για την αναχώρα έκθεσης και για τις αντίστοιχες ε, προδιαγραφές και τότε θα αποφασίσουμε ποια θέση θα κρατήσουμε. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε στην πορεία τα όσα αφορούν τον ορισμό της συμπεριφοράς των εταιριών και της υποχρέωσής τους για ενημέρωση για το πού λειτουργούν, πού συναλλάσσονται, ε, ώστε να μπορεί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, θα μπορούσαμε να περιμένουμε μέχρι ότου αποφασιστεί και αυτό το θέμα. Προχωράμε δηλαδή σε δύο παράλληλους δρόμους και μετά όταν θα έχουμε φτάσει σε συμπεράσματα, ελπίζω, όχι σε πολύ καιρό από σήμερα, χάρη στην βοήθεια που μας έδωσε και η Κομισιόν και η Ολλανδική Προεδρία, να μπορέσουμε ε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς με τη συμβολή των ε, σχεδόν και της Προεδρίας, ε, και θα προσπαθήσουμε βέβαια με την ε, απαραίτητη ταχύτητα να κάνουμε και τα όσα λείπουν για τα σημεία τα οποία σας ε, θύμισα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και έτσι θα περάσουμε στο θέμα των ερωτήσεων. Αλλά δεν βλέπω να τα κανείς το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν συνάδελφε Κόμφεράτη για το γεγονός ότι ήταν και συνοπτικότατος και θα περάσουμε λοιπόν στο σημείο υπερθμών 8 της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 7 θα το αναβάλουμε και θα περάσουμε στην παρουσίαση του έγγραφου του γράφω εργασία για τη μεταρρύθμιση των κανόνων περί πνευματική από τον Ζαν Καβαντά, συντονιστή τη ομάδα εργασία, τον οποίο και παρά θα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι και εγώ το πιο σύντομο δυνατόν γιατί ξέρω πως ε, τρέχει η ημερήσια διάταξη και για όσους δεν είναι ενημερωμένοι ο στόχος ήταν και αυτό το λέω για να έχετε μια πιο συγκεκριμένη άποψη και για όσους δεν συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για το, τη μεταρρύθμιση αυτή στα πνευματικά δικαιώματα. Να σας πω πως είναι ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο ούτε λαμβάνει θέση, ούτε υποστηρίζει κάτι συγκεκριμένο, απλώς κάνει μια απογραφή των όσων υπόθηκαν στην Επιτροπή που δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2014 με στόχο να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με όσο το δυνατόν περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη με όλους τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε η ομάδα εργασίας να μπορέσει να εξετάσει με τον κατάλληλο τρόπο και σε βάθος τις προκλήσεις που δημιουργούν αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και βεβαίως τώρα που μπαίνουμε στην ψηφιακή εποχή. Δεδομένου λοιπόν πως έχουμε αυτή την αναθεώρηση στα δικαιώματα αυτά, οι 15 πρώτοι μήνες αφιερώθηκαν αποκλειστικά σε αυτό το θέμα. Η ομάδα εργασίες από το Δεκέμβριο του 2014 συνεδριάζει. 109 επιρρογνώμονες ήρθαν και σε ακροάσεις κατά τη διάρκεια των 15 ε, συνεδριάσεις που κάναμε κάθε μήνα εκτός από τους θερινούς. Τι έχουμε στην έκθεσή μας. Η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει αρκετά ε, ζητήματα Καταρχήν έχουμε το δεύτερο τμήμα που έχει να κάνει με τις αμοιβέ και την αποζημίωση για τους ε, δημιουργούς και τους συγγραφείς. Δηλαδή ποιο είναι το σύστημα το οποίο θα υπολογίζει ποια είναι η αμοιβή που πρέπει να δοθεί σε ένα κόσμο ο είναι πολύ πιο ανοιχτός από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες. Το τρίτο έχει να κάνει με την εδαφικότητα ε, τις άδειες της ε, ε, γεωγραφικής εμβέλειας, όπως επίσης και τους περιορισμούς γεωγραφικούς. Μετά έχουμε το πώς επιβάλλονται αυτά μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το 5 έχει να κάνει με εξαιρέσεις και με περιορισμούς. Έχουμε το 6 που είναι η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. 7 η νομική βάση που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, για τα θέματα ε, copyright και μετά έχουμε τα υπόλοιπα, δεν θα σας πω ότι είναι ίσονο σημασία. αλλά για, επειδή είναι μικρότερο εύρος τα έχουμε εντάξει σε αυτό το 8ο κεφάλαιο. Μετά έχουμε τα συμπεράσματα και εκεί θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη γραμματεία η οποία έρχεται σε επαφή μαζί μας για να προετοιμάσει τις ακροάσεις και είναι πολύ ουδέτερη ε, η γραμματεία. Μιλάμε για μια τεχνική γνωμοδότηση και όχι πολιτική και γι' αυτό είχαμε θελήσει να έχουμε μια γκάμα πολύ μεγάλη εμπειρογνωμόνων. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, οι οποίοι συχνά έλαβαν μέρος στις συνεδριάσεις σε αυτή την Επιτροπή, επαναλαμβάνω μία φορά το μήνα. Και θα ήθελα να εκφράσω και τις ευχαριστίες μας ως Ευρωβουλευτές και ως μέλη αυτής Επιτροπής σε όλους τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που έρχονται για να μας φωτίσουν. Το έγγραφο είναι στη διάθεσή σας και θα κλείσω εκεί. Εάν θέλετε κάποια διευκρίνηση, ε, θα απαντήσω με χαρά, αλλά ήθελα να είμαι πολύ σύντομο γιατί όλα τα έχουμε ε, και σε κείμενο, οπότε δεν χρειάζεται εγώ να μακρηγορήσω. Ποιο θέλει το λόγο, κύριος Κέστερ. Äh, Ευχαριστώ πολύ για την εκθέση σα, κύριε Καβαντά. Πρέπει να σα πω πω η δουλειά που κάναμε μαζί για μένα ήταν ε, εξαιρετικά ε, επικοδομητική. Και η έκθεση ε, την οποία έχουμε ετοιμάσει είναι ένα καλό έγγραφο το οποίο θα μας βοηθήσει. Αυτό που είναι σημαντικό για το έγγραφο αυτό είναι ότι καταστήσει σαφές ότι μόνο η αγορά δεν μπορεί από μόνη της ε, να ρυθμίσει τα κοινωνικά δικαιώματα, θέματα πληρωμών με σωστό τρόπο. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάντα σωστό να εξετάζουμε σε τι βαθμό είναι δυνατόν σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πραγματική ιδιοκτησία, να την υπόψη και οι κοινωνικοί παράγοντε. Προκειμένου οι δημιουργοί πνευματικών ε, έργων πνευματική ιδιοκτησία να μπορούν να εξισωθούν με τους άλλους δημιουργού. γιατί βρίσκονται σε μια συγκριτικά δύναμη θέση τα άτομα αυτά. Πώ μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που παράγουν έργο τέτοιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, για παράδειγμα, στη Γερμανία εξετάζουμε το θέμα των ενώσεων, προκειμένου να μην παραμένει σε ατομικό επίπεδο, αλλά να υπάρχει και οργάνωση αρμόδια για τα άτομα αυτά και να εκπροσωπεί φυσικά τα δικαιώματά τους. Wir Uh, um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Καβαντά για την ε, παρουσίασή του και για τη γραμματεία που ε, συνέταξε αυτήν την ε, σύντομη έκθεση. Είναι μια καλή συνόψηση των διαφορών συζητήσεων που κάναμε και αναφέροντας σημαντικά σημεία θέλω να τονίσω ότι στην έκθεση λέει ότι Κάποιοι τομείς χρειάζεται να εξερευνηθούν περισσότερο, όπως α πούμε η σύνδεση ανάμεσα στις ε, ελεύθερε άδειες αλλά και τις διάφορες ενώσεις ε, που επιτρέπουν τη χρήση των διαφόρων ε, ελεύθερων αδειών αλλά και τη χρήση κάποιων πλάνων αποζημίωσης Ελπίζω πως θα βρούμε το χώρο ε, τον κατάλληλο σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις. Γενικότερα να πω ότι κάποιες φορές συζητήσαμε, είχαμε το πρόβλημα μάλλον ότι είναι σχετικά δύσκολο να καλέσουμε ε, ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς πυρογνώμονες για, απλά και μόνο για θέματα πρακτικά έχουν δυσκολία να φύγουν από τις ε, εργασίες τους ή να πληρώσουν για το ταξίδι θα μπορούσαμε ίσως λοιπόν να έχουμε περισσότερες γραπτές εμπειρογνωμοσύνες ή να γίνουν συζητήσεις στην Επιτροπή μας που μπορούμε να καλέσουμε τους ειδικού. Οι απόψεις ανεξάρτητων πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων είναι νομίζω πολύ σημαντικές. Ιδιαίτερα όταν ασχολούμαστε με το τομέα των, ε, ιδιωτικ... της πνευματικής Ο εισηγητής μας ο κ. Καβαντάς θα είστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί θα το πω πολύ γρήγορα, γιατί οι συνάδελφοι και οι παρατηρήσει του είναι προφανεί. Οπότε τη σημειώνω βεβαίω Να κλείσω από εσά, κυρία Ρεντά. Σα ευχαριστώ για τι ευχαριστίε σα, για όλου όσου εργάστηκαν ε, για αυτό το θέμα, όχι μόνο δηλαδή για του ευρωβουλευτέ. Και επίση να πω ότι σημειώνω από πολύ προσοχή όσα μόλι είπατε. Και εγώ όπως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστερ για τη δουλειά που κάνατε σε αυτήν την επιτροπή. Είστε μονίμως παρόν, είστε πολύ ενήμερος. Ε, για τα θέματα. Η ιδιαιτερότητα της Ευρώπης σε σχέση με τις άλλες υπήρους όσον αφορά την ψηφιακή ε, τεχνολογία αλλά και τα θέματα περιεχομένου, δηλαδή αυτών που τροφοδοτούν τη ψηφιακή τεχνολογία, είναι ακριβώς ε, μια ισορροπία που η ισορροπία των θεμάτων αυτών τίθεται με μεγαλύτερη ακρίβεια γιατί όλοι Κάποιες φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα δύο συστήματα προμήθειας και χρήσης. Ε, και για, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι βλέπουμε πολύ καλά ότι οι ανάγκε τη ψηφικής βιομηχανία αλλά και της ε, καλλιτεχνική βιομηχανία δεν είναι αντίπαλοι. Αντίθετα, είναι δύο στοιχεία μιας η ζωντανή αλυσίδα που τροφοδοτεί την πολιτιστική μας ε, ε, ταυτότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο 10 της ημερησίας διάταξης. Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην ιστορική ναυσιπλοεία. Να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Μπερσέγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή που έχω να σας υπενθυμίσω ότι μετά τις πλημμύρες που στη Γαλλία που έπλεξαν τη Γαλλία, όλοι στις διάφορες επιχειρήσεις ε, που έχουν τα τουριστικά πλοιάρια στο Παρίσι και που ε, ε, και οι οποίοι εξυπηρετούν τουλάχιστον 20.000 τουρίστες την ημέρα, ε, πρέπει να σας πω πως η σκέψη μας είναι μαζί τους, γιατί ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες οικονομικά ε, έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Τώρα, νομίζω ότι για τη γνωμοδότηση τη δική μας είναι μια γνωμοδότηση για το σχέδιο οδηγίας για την αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματικών στην εσωτερική ναυσιπλοεία και να σας πω πως μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους εμπλεκόμενους στις ενιάλειες μεταφορές να σας πω πως δεν είχαμε καμία βασική ή μεγάλη αντίδραση στα όσα προσπαθούν να κάνουμε και βεβαίως η μεγαλη αντιδραση στα οσα προσπαθουν να κανουμε και βεβαιως η κατάργηση των δύο προηγούμενων ε, οδηγιών, του 91 και του 96, έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε μόνο ε, τους ε, καπετάνιους αυτών των πλοίων και δεν συμπεριλάμβανε και τον Ρήνο. Οπότε εδώ θα συμπεριλάβουμε και όλα τα πληρώματα, κάτω και από το βαθμό δηλαδή του πλειάρχου και την περίπτωση του ρήνου, για όσους δηλαδή μεταφέρουν επιβάτες ε, στα ποτάμια στην Ευρώπη. Εδώ δεν καλύπτουμε βέβαια τα σκάφη αναψυχής, μόνο ε, όσους ε, κάνουν μεταφορά επιβατών. Δίνονται και κάποιες εξαιρέσεις για κάποιες πλωτές οδούς ε, που δεν ε, καλύπτουν καμία διασυνοριακή ε, μεταφορά. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να προκρίνουμε αυτή την δυνατότητα τουρισμού γιατί αυτή η μεταφορά ανταποκρίνεται απολύτως ε, στις τρεις, στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό επίπεδο. Είναι ανταγωνιστικές οι, τιμές σε σχέση ε, με τις ε, οδικές μεταφορές. Δεν έχει πολλές εκπομπές αερίου θερμοκηπίων και επίσης δεν ε, είναι ε, ενεργοβόρα. Δηλαδή ε, ένας τόνος εμπορευμάτων που χρειάζεται για να μεταφερθεί ένα τόνο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, εάν μεταφερθεί με φορτηγά, θα χρειαστεί μόνο το ίμιση αν μεταφερθεί πλωτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά για τους γερμηνείς Με συγχωρείτε μου είχατε πει ότι πρέπει να το πω γρήγορα. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν προκαλεί πολλά ατυχήματα και δίνει μεγάλες δυνατότητες ε, ανάπτυξης στις ροές, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πολλές καινούργιες νέες θέσεις απασχόλησης, κυρίως στα ε, λιμάνια. Και είναι ε, μια, ένας κλάδος ο οποίος χρειάζεται χέρια, 3.600 θέσεις αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, με πολλές προοπτικές για το, ε, για το μέλλον και έχουμε επίσης ε, και τον Σικουάνο που θα μπορούσαμε να ε, πολλαπλασιάσουμε επί πέντε τις μεταφορές και στον Ρήνο 8 ή 9 φορές περισσότερες θα μπορούσαν να γίνονται αρκεί να είχαμε την απαραίτητη ε, κατασκευαστική δραστηριότητα που θα μας επέτρεπε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Να δούμε λοιπόν και ποιες είναι οι απαιτήσει σε επίπεδο αναγνώριση και ποιες είναι οι τοπικές ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η δυνατότητα να εισάγουμε κάποιες ελάχιστες απαιτήσει για τα επαγγελματικά ε, προσόντα, για τους κατόχους και για τους πλειάρχους αυτών των σκαφών είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Θα πρέπει αυτές οι εσωτερικές πλωτοί όταν είναι διασυνοριακής φύσης, να μπορούν να διατηρήσουν παράλληλα τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά, τα συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά που του ταυτοποιούν. Και για το λόγο αυτό πιστεύω πως θα έπρεπε να αφήσουμε ανοιχτή τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν και κάποιες εξαιρήσει, όπως για παράδειγμα για τις ε, ε, περιπατητικές δραστηριότητες ή ε, για τον τουρισμό στα ποτάμια ε, που συνήθως ε, ασκείται από πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Εγώ προσπάθησα να εμπνευστώ από την οδηγία που αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε για τις τεχνικές προδιαγραφές για τα σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοείας και να σας πω πως οι τροπολογίες που προτάθηκαν έχουν να κάνουν με τα προσόντα, τα επαγγελματικά, για το σύνολο των κρατών μελών που έχουν πει πως για τη συμμόρφωση ε, θα ε, εξαντλήσουν την προθεσμία έτσι ώστε να μην επιβάλλουν ε, κυρώσεις σε αυτή την αγορά δημιουργώντας μία σπάνιση των ανθρώπινων πόρων και είπαμε μια μεταβατική απερίοδος μεγαλύτερη που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σιγά σιγά να συμμορφωθούν με τις απαιτήσει που υπάρχει στην οδηγία και στα παραρτήματά της. Και γι' αυτό στην τροπολογία 10 θελήσαμε να μεταφέρουμε ε, στα πέντε έτη τη μεταβατική περίοδο και να μην παραμείνουμε στα τρία έτη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην τροπολογία 11 προτείνουμε η οδηγία να μιλά μόνο για τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοιου είδους εσωτερικές πλωτές οδούς, σαν αυτές που έχουμε στο άρθρο 3. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι και με μεγάλη χαρά θα ανταλλάξω απόψεις μαζί σας ε, για όλα τα στοιχεία αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Thank you very much. Any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 Uh, the Commission wishes to take the floor. Okay, you, you have it. Thank you very much, Mr. Chairman. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Ιστολογίτης και είμαι επικεφαλής της μονάδας που ασχολείται με τα θέματα ιστορικής πλόγησης ιστορικών πλωτών οδών. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εισήγηση σε ένα περίπλοκο θέμα. Μέσα σε πέντε παραγράφους μας δώσατε μια πολύ καλή ιδέα για το τι είναι αυτό το θέμα και τι προσπαθεί να κάνει αυτή η οδηγία. Θέλω να συνοψίσω με δύο φράσεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις εσωτερικές πλωτές Πρώτον, δεν έχουμε νέο αίμα. Έχουμε πρόβλημα με την πυραμίδα των ηλικιών που είναι πολύ πιο έντονο και πολύ πιο βαριά είναι η πυραμίδα στο πάνω-πάνω μέρο της και πολύ ελαφριά κάτω-κάτω γιατί ο κόσμος, τα νέα παιδιά δεν βλέπουν προοπτικές και δεύτερον υπάρχει και μια δομική ανισορροπία ανάμεσα στην ζήτηση για πληρώματα και την προσφορά. Η ζήτηση είναι στην περιοχή του Ρήνου, όπου υπάρχει το 70% της κυκλοφορίας, αλλά δυστυχώς η προσφορά προέρχεται από άλλα μέρη της Ευρώπης. Γι' αυτό τον λόγο θέλουμε να προτείνουμε έναν ενιαίο χώρο όπου όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το επάγγελμα, να μπορούν να το ασκήσουν. Είτε ξεκινούν ως απλοί ναυτικοί, είτε φτάνουν μέχρι το καπετάνιο. Ε, προσφέρουμε δηλαδή μια σταδιοδρομία ώστε να μπορούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα οπουδήποτε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το κύριο πλανέκτημα αυτής της πρότασης. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αυτές την εισηγήτρια με συγχωρείτε, για αυτές τις τροπολογίες που είναι πολύ αντικειμενικές όσον αφορά τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, αλλά έχω ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω να θίξω. Και αυτό είναι το εξή. Όταν στην τεχνική οδηγία που έχει θεωρηθεί παράδειγμα γίνεται διάκριση ανάμεσα σε ε, ζώνες πλοήγησης, έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές συνθήκες των υδάτων. Η ζώνη 1, 2, 3 και 4 και μετά έχουμε τη ζώνη του Ρήνου που είναι πολύ διαφορετική. Έχει πολύ διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα σκάφη κατασκευάζονται διαφορετικά γιατί πρέπει να έχουν διαφορετικές αντοχές. Ενώ τα πλοία που πηγαίνουν στην, ε, στη ζώνη 4 πρέπει να έχουν πιο ε, γέρη κατασκευή. όμως δεν είναι οι άνθρωποι που πρέπει να ενδιαφέρουν. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τις ίδιες ικανότητες τι ίδιες δεξιότητε, όπου και αν πρέπει να ε, εργαστούν. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε ένα ομοιόμορφο σύστημα ανεξάρτητα από τις ζώνες. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα αναζώνη, αυτό σημαίνει ότι ένα επαγγελματία οδηγό που έχει πάρει τη δίπλωμα οδήγησή του στην Ολλανδία δεν θα μπορούσε να, ε, να οδηγήσει στην Αυστρία, στην ε, Ελβετία, γιατί εκεί έχει βουνά. Αλλά δεν είναι αυτό ο τρόπο για να δημιουργήσουμε μια αναγορά για τους επαγγελματίες που θέλουν να μπορούν να ασκήσουν το επαγγελμά τους οπουδήποτε στην Ευρώπη. Για αυτό το συγκεκριμένο αυτό λόγο λοιπόν είπαμε ότι το χάλιβας και το πάχος του χάλιβα για τα σκάφη μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά οι ναυτικές δεξιότητες πληρωμάτων ε, και εργαζόμενων εκεί είναι ε, οι ίδιες. Για κάποιον που εργάζεται ας πούμε, στο κανάλι του ΜΙΔΙ που δεν μπορεί ή δεν θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή πλοήγηση, προβλέπουμε εθνικέ εξαιρέσει. Αλλά για όλους τους άλλους είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό παντού στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό έχουμε πρόβλημα με αυτές τις τροπολογίες που και πάλι προσπαθούν να, αποκαταστήσουν να, να, να εισάγουν μια, έναν κατακαιρματισμό που θα είναι κατά της κινητικότητας των εργαζομένων στο τομέα. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα αυτή την έκθεση. Πρόκειται για μια πρόταση, όπως σας είπα, που στόχο έχει να ενοποιηθεί αυτή η κατακαιρματισμένη σήμερα κατάσταση. Δύο σύντομες παρατηρήσεις ακόμα όσον αφορά την προθεσμία για τη μεταγραφή. Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, δεν έχουμε πρόβλημα με μακρύτερη περίοδο μεταγραφής. Ωστόσο έτσι θα καθυστερούσαν τα ωφέλη για όσους επιθυμούν να μπουν σε αυτό το νέο σύστημα. Πρέπει να τα σταθμίσουμε λοιπόν αυτά. Και τέλος, για την εφαρμογή, της εφαρμοστικές και τις συμπράξεις είναι πιο θεσμικό το θέμα, δεν χρειάζεται να μπω ε, με λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα τώρα. Συνοψίζοντας λοιπόν να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά Θέλω να δούμε αν είναι τελικά επιθυμητό να σκεφτούμε εάν είναι επιθυμητό να συνεχίσουμε με τον κατακαιρματισμό και να εισάγουμε και περισσότερο κιόλα. Ε, ε, και μήπω είναι καλύτερα να προχωρήσουμε προ ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σχολιάσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, very... ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Θέλει η συγκεκριμένη να σχολιάσει ή να Είχα καταλάβει πως υπάρχουν ζώνες και καταλαβαίνω πως αν είναι κανείς οδηγός ε, τρένου ε, δεν μπορεί να γυρίσει να οδηγεί το τρένο στο Βέλγιο γιατί είναι διαφορετικές οι ράγες για παράδειγμα, είναι διαφορετικά τα προσόντα που χρειάζεται αλλά ένα πλοίο το οποίο το νοικιάζουμε σε κάποιους εκδρομείς ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει το ίδιο πρόβλημα. Είπαμε, εθνικές ε, εξαιρέσεις. Νομίζω ότι με αυτό το καλύπτουμε. Πάντως για τα πέντε χρόνια θα επιμείνω. Ξέρω τι σημαίνει για τον κλάδο. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι λοιπόν ολοκληρώσουμε και το σημείο αυτό, το υπαριθμό 10 στην ημερήσια διάταξη και ας πάμε, ας επανέλθουμε στο σημείο 7 Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ετήσια έκθεση για το 2014. Τώρα η κυρία Χάουταλα, η εισηγητρία. Ευχαριστώ, πρόεδρε. 63 είναι οι τροπολογίε οι οποίε λάβαμε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες εξ αυτών. Συνολικά θα έλεγα ότι η ιδιαίτερη έμφαση της φετινής έκθεσης ε, ήταν ευπρόσδεκτη με κάποιες αποχρώσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην ε, υλοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου στις ε, χώρες της συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οποίες έχει εταιρικό καθεστώς ε, συνεργασίας η Ένωση. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι πιο πολλοί εξημών θέλουν να υπογραμμίσουν ότι χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρακτικά αυτά προγράμματα. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις αντικαθιστά πλήρω τις διαδικασίες επί παραβάση. Επί του παρόντος, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίε για να κατανοήσουμε γιατί σε κάποιε περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακόπτει τι ε, διαδικασίε και γιατί σε κάποιε άλλε θα συνεχίζει. Κάποια άλλα θέματα σε ό,τι αφορά το θέμα της επικουρικότητας. Μας απασχολεί στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα ωστόσο, μάλλον επειδή δεν είναι τη αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα τα θέματα αυτά, να μην τα θέσουμε εδώ. Επίσης, το ECR κατάθεσε κάποιε τροπολογίε για τον κανονισμό για την ανοιχτή, αποδοτική και διαφανή διοίκηση της Ένωσης αλλά είναι διτεθμένοι να τις αποσύρουν, γιατί δεν συνάδευτε με το γενικότερο στόχο της νομοθεσίας. Χαίρομαι που είναι εδώ και ο κύριο Σβίφκα και χαίρομαι πάρα πολύ που κατέθεσε και τροπολογία για το gold plating αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα και τον απασχολείται το θέμα αυτό και πραγματικά συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες που έχετε θέσει για το θέμα αυτό του gold plating. Το 14 θα θέλαμε να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις τις εφαρμοστικές είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή και κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή συνολικά. Επίσης, αναμένουμε γνωμοδοτήσεις από 8 επιτροπές. Τις τρεις τις έχουμε ήδη λάβει. Οι νομοθετικές επιτροπές της ε, του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Αναφορών που έχει ιδιαίτερο συμφέρον από πλευρά ε, των συμφέροντων των πολιτών να παρακολουθεί θέματα εφαρμογή ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα ήθελα να δείξω μια ειδική τροπολογία που λάβαμε από την νομοδότηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Μια έκκληση για ένα πιο διαρθρωμένο τρόπο παρακολούθησης εδώ στο Κοινοβούλιο των ε, υποθέσεων αυτών. Αυτό θεωρώ ότι αποτυπώνει ιδέες και προτάσεις που ε, έχω ακούσει σε διάφορες περιστάσεις τελευταία. Και έχω ακούσει σε διάφορες περιστάσεις ότι θα έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει συντονιστικό ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή δουλειά από όλες τις Επιτροπές τελευταίο λοιπόν σημείο της γνωμοδότησης της Επιτροπής ΕΚΟΝ αναφέρει ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ υποστηρίζει την δημιουργία διαρθρωμένης δομής στα σκόλπους του Κοινοβουλίου για την ανάλυση των ζητημάτων μη συμμόρφωσης με τρόπο που θα είναι συγκεκριμένος αναχώρα και θα λαμβάνει υπόψη ότι οι μόνιμες επιτροπές με αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα ανάλογα με τον τομέα αρμοδιοτήτων. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, τη συζήτησα με τον εισηγητή, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να υπάρξει υποεπιτροπή για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και αυτό κυκλοφορεί σαν ιδέα. Και ξέρω ότι η διάσκεψη των Προέδρων Θέλω να δραματίσει ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ότι εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή για να κάνουμε το συντανισμό και θα πρέπει αυτό να γίνει με πιο τρόπο. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές. Ελπίζω λοιπόν να σας ε, αρκούν τα στοιχεία αυτά. Προφανώς θα ψάξω και θα βρω καλούς συμβασμούς ε, στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι οι τροπολογίες για θέματα επικουρικότητας δεν έχουν να κάνουν με την έκταση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κάφμαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια ζητήματα θα ήθελα να θίξω, γιατί υπάρχουν στροπολογίες, κάποια ζητήματα σε, τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Η 14 και 15 τροπολογία, για παράδειγμα όπου μιλάμε για καλύτερη εξάντου προετοιμασία των κρατών μελών με πίνακες αντιστοιχεία. Στο ζήτημα επίσης ε, συζητιέται επιμακρών για τη δική μου έκθεση σε ό,τι αφορά το gold plating, τον νομοθετικό υπερθεματισμό. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μία σωστή έξπος σήμανση από πλευρά των κρατών μελών που δεν σχετίζεται απαραίτητα με την κοινωτική ρύθμιση. Επίσης, τροπολογίες που επικεντρώνοντας το ρόλο του Κοινοβουλίου, στην ενίσχυση του ρόλου αυτού και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μετά από όσα μας είπε και η κυρία το θέμα της γνωμοδότησης σε ό,τι αφορά και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ένα σημείο επίσης θα ήθελα ρητά να υποστηρίξουν την εισηγήτρια το θέμα της, ε, των τροπολογιών που έγιναν για την επικουρικότητα. Με παραξένεψε ιδιαίτερος. Πολύ σημαντική η επικουρικότητα και προφανώς και συζητιέται επισταμένως. Αλλά εδώ, το αντικείμενο της έκθεσης είναι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μιλάμε για θέματα ελέγχου επικουρικότητας. Θα έλεγα λοιπόν να το να τα διαγράψουμε εντελώ τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την επικουρικότητα. Έχουμε άλλωστε και την έκθεση ελέγχου επικουρικότητα του 2015 και να τα κοιτάξουμε αυτά. Και θα περιμένουμε και τις συμβαστικέ προτάσεις τη ηγήτριας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Ε, ευχαριστώ, κυρία Σβιεύκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω και την κυρία Χάουτουλα και εγώ για την έκθεση αυτή και για την παρουσίαση των ε, τροπολογιών. Πολλέ, πολλέ, δεν λέμε, αλλά να μην ε, μα αποθαρρύνει αυτό, έχουμε δει και χειρότερα. Θα τα καταφέρουμε. Πόσο μάλλον που μα είπε και η συγγήτρια ότι ένα μεγάλο κύμα των τροπολογιών δεν έχει να κάνει με την έκθεση κιόλα. Και εγώ θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή προσέγγιση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και σε ό,τι αφορά το gold plating, το νομοθετικό υπερθεματισμό. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο μας απασχολείται και χρόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η έκθεση αυτή μπορεί να έχει επίδραση με μόχλευση για τη δουλειά μας εδώ. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση, αλλά τα εργαλεία, η άμεση εφαρμογή στα κρατή μέλη, αυτό βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή έχει επισκόπηση υπέρ του θέματος, αυτά που συμβαίνουν με την οδηγία, τα κρατη και διάφορες ομάδες κρατών που δεν εφαρμόζουν διατάξεις. Μας κάνει την ε, ζωή δύσκολη, γιατί πραγματικά κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως είναι καλό και φατικό, αποδεικνύεται υπερβολικά δύσκολο. Και πραγματικά αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει. Μοιραία. Άρα πλέον αυτό θα πρέπει να γίνει επειδή το θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, το θέμα είναι και τι θέλει και κάθε κράτος. Ε, υπάρχει δυνατότητα λοιπόν και περιθώρια ερμηνείας και αυτό μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ένα καλό συμβιβασμό όπως σας είπα και σε τελική ανάλυση να πετύχουμε μια καλή έκθεση από πλευρά της κυρίας Χάουτουλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Δεν ζητά κανείς άλλος το λόγο και ως εκ τούτου μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει το 12 και το 9. Μήπως θα μπορούσαμε να το αναβάλουμε. Να πάμε στο 28. 28. Ανταλλαγή δηλαδή απόψε σε ό,τι αφορά τι δηλώσει οικονομικών συμφερόντων των επιτρόπων κατά την κυρία Θαναμέ. Πασκαλουριά, εισηγήτρια, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσπαθήσω κι εγώ να επιτρέψω σε αυτή την επιτροπή να κερδίσει χρόνο, γιατί νομίζω πως με αυτή την ε, πρώτη παράμβαση για τις ε, εργασίες που έχουν γίνει και από τη Γραμματεία και από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και για τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια έχουμε κατά τη γνώμη μου μια θέση στο ιστορικό του Κοινοβουλίου που μπορεί να είναι απολύτως συνενετική. Δεν θα επανέλθω στις δυσκολίες που είχαμε αρχικά για να δούμε ποιους είναι ο ρόλος της Επιτροπής μας, αυτή την εξέταση των δηλώσεων των οικονομικών συμφερόντων που θα πρέπει να καταθέσουν οι Επίτροποι, εμείς κάναμε τη συζήτηση, βρήκαμε ε, πως πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ έκανε τη δουλειά της και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα αυτό για να προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε τη θέση αυτή στα πλαίσια της Επιτροπής μεταξύ του θέματος των δηλώσεων οικονομικών οικογενειακών συμφορέντων με την ευρύτερη έννοια που για έναν επίτροπο ε, θα σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο φάκελο δεν θα μπορεί να τον αναλάβει και να περάσουμε σε μια αφετηρία στη στιγμή του διορισμού όπου έχουμε μόνο αυτή τη δήλωση την προσωπική των οικονομικών συμφερόντων Euh, Και το οποίο σημαίνει πως η θέση που λαμβάνουν κάποιοι επίτροποι δεν είναι απαραίτητο ή καλύτερη, χωρίς αυτό να θίγει την καταλληλότητα ε, του επιτρόπου που μπορεί να είναι πραγματικά ε, εξαιρετικών ικανοτήτων. Άρα λοιπόν υπάρχει το θέμα του να προλαμβάνονται οποιαδήποτε τέτοια συγκρούσει συμφερόντων πριν το διορισμό, γιατί δεν είναι ούτε ο ρόλο ο δικό μα να χρειάζεται να αποφασίσουμε εμείς για το ποια είναι η αρμοδιότητα των επιτρόπων, ούτε, και επιμένω εδώ, και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι για το οποίο κατηγορήθηκα σε κάποιο βαθμό στην αρχή και λυπάμαι γιατί ίσως δεν εκφράστηκα καλά. Δεν είμαστε δικαστήριο και δεν είμαστε εδώ εμείς για να δικάσουμε τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε εδώ για να εξετάσουμε απλά αν υπάρχει ή όχι κίνδυνος σύγκρουσης εμφορώντων σε συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό θα κάνουμε. Είμαι πεπισμένος πως μπορούμε να το κάνουμε καλά. Και είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας για οποιονδήποτε συνάδελφο που ήδη θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Πάντως θέλω να σας καθησυχάσω δεν είναι για μένα και καθόλου δεν είναι το πνεύμα αυτό το οποίο με εμπνέει να ακολουθήσω μια λογική εισαγγελία ή δικαστηρίου εναντίον οποιοδήποτε, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εκτό αυτή. Και θέλω εδώ να επιμείνω. Ε, thank you, Mr. Merci, Président. Très rapidement, je... Κύριος Okay. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω κι εγώ, έχοντας ακούσει τον κύριο Ντυρό, πώς αντιμετωπίσαμε δύο εμπόδια την τελευταία φορά που έγινε η συζήτηση με τους επιτρόπους στην αρχή της αιτίας, μας ζητήθηκε να ευλογήσουμε την πρόταση που κάνουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και συμφωνώ απολύτως με τα όσα εκφράζατε, αλλά πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τα μέσα για να εξετάσουμε την ειλικρίνεια των δηλέσεων που μας υποβάλλονται εμείς χρειάστηκε να εμπιστευτούμε τα όσα ήταν καταγεγραμμένα στις δηλώσεις αυτές. Και σε δύο περιπτώσεις τα 10 χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια με δύο διαφορετικούς επιτρόπους σε διαφορετικές θέσεις βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση και επίσης πρέπει να σας πω πως στηρίζω πάρα πολύ τα όσα είπε ο κύριος Ντυρό. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, δεν είμαστε ανακριτές δεν μπορούμε να εξετάσουμε την ειλικρίνεια των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφεύγονται τέτοιου είδου συγκρότηση συμφερόντων. Γιατί ε, καταλαβαίνετε ε, πόσο αυτά ε, φαίνονται άσχημα εκτός του οίκου μα. Θυμόστε τι έγινε το 2014 με το διορισμό τότε συγκεκριμένου επιτρόπου. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Uh, Η κυρία Ρέγνερ. Ε, ε, Δεν θα μακρηγορήσω, ευχαριστώ. Νομίζω ότι και ο κύριο Ντυρό και ο κύριο Καβαντά τα παρουσίασαν όλα πολύ συνοπτικά και σωστά σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήριες γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι σχετικέ. Παρατηρήσει. Τα εξέτασα όλα αυτά και θεωρώ ότι αποτελούν ένα πολύ καλό πλαίσιο για να γίνουν οι εργασίες μας και να συνεχιστούν οι συζητήσεις μας. Ασφαλώ. Και βεβαίω δεν είμαστε ερευνητική επιτροπή. Ούτε δικαστήριο. Αλλά η επιτική γωνία μας δεν είναι αμυγός από την πλευρά των ε, διεδικαστικών σφαλμάτων ή όχι. Όχι, χρειαζόμαστε λίγο πιο ευρύ βλέμμα και οπτική γωνία. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Ντουράν, σύμφωνα με τα σχόλια που κάνατε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν ζητάει το λόγο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε και το 28. Πάμε στο 13 και 15. Έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων των εκτελεστικών μέτρων. Και το λόγο παίρνει η κυρία Κάφμαν, η εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είμαστε σύντομες. Σύντομοι. Από πλευρά τη δικιά μα ε, και των συναδέλφων δεν ε, υπάρχουν ε, οποιασδήποτε παρατηρήσει. Θεωρούμε ότι όλα ήταν όπως έπρεπε. Όλα εντάξει. Yes, I think that Mrs. Kaufman should... Νομίζω ότι η κυρία Κάφμαν νομίζω πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα και παράδειγμα για όλους τους επόμενους ομιλητές. Πολύ σας ευχαριστούμε και τώρα συνεχίζουμε αλλά και κλεισμένον το θηρεών. Όποιος λοιπόν δεν δικαιούται να παρευρεθεί σε συνεδρίαση και κλεισμένο βαθρών, παρακαλώ να εξέλθει τις αίθουσες.